Ladies and gentlemen, please be seated. και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. So once again, ladies and gentlemen, please be Καθίστε, παρακαλώ. Ελπίζω να υπάρχουν θέσεις ακόμα. συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα να καλωσορίσω τον κύριο Ζωζέ Μπορέλ, υποψήφιο για την θέση της, του είπατε για τα εξωτερικά και την αμυντική ασφαλείας. Καλώς ήρθατε λοιπόν κύριε Μπορέλ. Χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ πέρα απόψε γιατί πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία για διάλογο και το πρώτο βήμα προς μια επικοδομητική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βεβαίως ε, μας γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και δεν έχω καμία αμφιβολία πως θέλετε να έχουμε στενές σχέσεις και επαφές ε, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο μέλλον. Θα ήθελα να υπενθυμίσω συναδέλφους πως ο στόχος αυτής της ακρόασης είναι το Κοινοβούλιο να αξιολογήσει τον υποψήφιο επίτροπο με βάση την γενική του ικανότητα, την προσήλωσή του στα ευρωπαϊκά ιδανικά και την προσωπική του ανεξαρτησία. Επίσης, μας δίνεται η δυνατότητα να αξιολογηθεί η γνώση του υποψηφίου επιτρόπου στο χαρτοφυλάκιό του και οι ικανότητες επικοινωνίας. Κυρίες και κύριοι, στις 25 ε, Σεπτεμβρίου λάβαμε τις απαντήσεις του κυρίου Μπορέλ. Τι έχουμε μοιράσει σε βουλευτές σε όλες τις γλώσσες και επίσης δημοσιεύτηκαν στην σελίδα του Κοινοβουλίου. Τώρα θα ήθελα σύντομα να περιγράψω το πώς ε, θα διεξαχθεί αυτή η ακρόαση σύμφωνα με τους ε, κανόνες του Κοινοβουλίου για να έχουν όλοι οι υποψήφοι επίτροποι την ευκαιρία να παρουσιάσουν αυτούς και απόψεις. Πρώτα απ' όλα θα υπάρξει μια αρχική δήλωση που δεν θα διαρκέσει πάνω από 15 λεπτά μετά από την εισαγωγή αυτή. Θα υπάρχει ο χρόνος για 25 ερωτήσεις από τους βουλευτές. Στον πρώτο γύρο θα έχουμε τις ερωτήσεις ε, των ε, ομιλητών των πολιτικών ομάδων και μετά τις ερωτήσεις 18 βουλευτών σύμφωνα με την ποσόστοση ε, που γίνεται μεταξύ των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων. Τα 5 λεπτά θα πάνε ως εξής. Κάθε βουλευτής έχει ένα λεπτό για να κάνει την ερώτηση του ή της και μετά ακολουθεί μια απάντηση δύο λεπτών από τον υποψήφιο επίτροπο. Μετά, αν απαιτηθεί, υπάρχει δυνατότητα να γίνει άλλη μια ερώτηση, το πολύ ενός λεπτού και ο υποψήφιος επίτροπος μετά θα δώσει μια μονόλεπτη απάντηση στην ερώτηση αυτή. Να υπενθυμίσω συναδέλφους πως η δεύτερη ερώτηση πρέπει να έχει κάποια σχέση με την απάντηση στην πρώτη ερώτηση και ε, δεν θα αφορά άλλα ζητήματα στο τέλος της ακρόασης. Ο υποψήφιος επίτροπος θα έχει 5 λεπτά για να κάνει μια δήλωση. Ο συνολικός χρόνος ε, της ακρόασης είναι 3 ώρες αυστηρά. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να παραμείνετε εντός του χρόνου. Εάν μιλήσετε περισσότερο, σημαίνει ότι αφαιρείτε το χρόνο από κάποιον συνάδελφο. Γι' αυτό έχω αυτό το σφυράκι. Δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω, αλλά σας προειδοποιώ. Εάν μιλήσετε περισσότερο, θα χτυπήσω το σφυράκι και όταν το χτυπήσω δύο φορές σας αφαιρείτε το μικρόφωνο. Τέλος, διερμηνία έχουμε σε όλες τις γλώσσες και η συνεδρίαση μεταδίδεται στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου και θα υπάρχει και η δυνατότητα να την δείτε μαγνητοσκοπημένη. Πριν δώσω τον λόγο, θα ήθελα να τονίσω την σημασία που έχει αυτή η ακρόαση για έναν αποτελεσματικό διάλογο μεταξύ του ΙΠΑ του εκπροσώπου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια στιγμή κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις αλλά μπορεί να παίξει και έναν σημαντικό ρόλο στην ε, προώθηση λύσεων για τόσα σημαντικά ζητήματα και είναι σημαντικό να τονίσουμε την κοινοβουλευτική διάσταση της εξωτερικής ε, δράσης ε, και την διοργανική συνεργασία. Αυτά από εμένα. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, έχετε τώρα τον λόγο. Για 15 λεπτά ακριβώς έχετε τον λόγο. Αγαπητοί βουλευτές, με χαρά μου ξαναγυρίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με κάθε ταπεινότητα ε, αισθάνομαι ότι είναι τιμή για μένα για όλες αυτές τις ε, αρμοδιότητες οποίες θα αναλάβω και αναγνωρίζω το πόσο σημαντική είναι η Συμβουλή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαμόρφωση της εξωτερική πολιτικής της Ένωσης και την προστιθέμενη ε, αξία ε, που ε, συμβάλλατε στην υπόθεση της Ουκρανίας και μία αρμοδιότητά μας θα είναι να ενημερώνουμε, να διαβουλευόμαστε ε, και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το ότι λαμβάνεται υπόψη γνώμη του Κοινοβουλίου. Θέλω μια ισχυρή εξωτερική πολιτική της Ένωσης και αυτό απαιτεί ε, δημοκρατική νομιμότητα. Και σε αυτή την ε, αρχική μου δήλωση θέλω να δούμε ενοιολογικά τα θέματα και όχι γεωγραφικά για την οικονομία της συζητήσεως. Αλλά θα ήθελα από την αρχή να σας ξεκαθαρίσω ότι προτίθεμαι να προχωρήσω σε μεταρρυθμίσεις και σε ε, διαδικασία ολοκλήρωσης στα Δυτικά Βαλκάνια για να βοηθήσω στην δημοκρατία και θέλω να ε, ε, αποκατασταθεί η ενότητα της χώρας στην Ουκρανία, επίσης και στα νότια σύνορα της χώρας, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να έχουμε μια συνολική στρατηγική σε σχέση με την Αφρική. Θα πρέπει να επεξεργαστούμε τις σχέσεις μας με την ε, Ασία και να αναβαθμίσουμε τη συνεργασία με την ε, Αμερική και τις υπερατλαντικές σχέσεις όμως, όπως είπαμε, πρόσφατα με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Πομπέο. Θα πρέπει να τις ε, επανακαθορίσουμε τις σχέσεις μας με τις ε, υπαπέραν αυτών, να δούμε επίσης πώς είναι δυνατόν ε, χέρι-χέρι να προχωρήσουμε για δημοκρατία, για ανθρώπινα δικαιώματα στην εποχή των τόσων προκλήσεων. Πρώτα-πρώτα να σας πω συνολικά τι όραμα έχω. Κύριοι βουλευτές, Κύριε Πρόεδρε, σύντομα θα έχουμε την 30η επέτειο της ε, πτώσης του τείχους του Βερολίνου. Επρόκειτο για θρίαμβο της ελευθερίας. Έτσι και ήταν εφικτή η επανένωση της δημοκρατίας Τη ελευθερια ετσι και ηταν εφικτη η επανενωση τη δημοκρατιας δημοκρατία στην ε, Ευρώπη. Ε, έφερε όμω αυτό το γεγονό, διάφορε άλλε προκλήσει οδηγηθήκαμε έτσι στο ευρώ, στην διεύρυνση και σε μια κοινή εξωτερική πολιτική. Και Τότε υπηρέτησα το κοινοβούλιο και εγώ, αλλά από τότε έχουν γίνει εντυπωσιακέ θεματικέ αλλαγές παντού. Και προς το χειρότερο, πολύ χειρότερο. Έχουμε το μεταναστευτικό, το προσφυγικό, αστάθεια στη γειτονιά μας, έχουμε τις κυβερνοαπειλέ και επομένω βλέπουμε ότι έχουμε την λογική ε, της ε, ισχύω. Τα πράγματα δεν είναι δίκαια, τα πράγματα είναι απρόβλεπτα. Ε, και οδηγούν σε συγκρούσεις. Power politics το λέμε, ότι δηλαδή δεν ισχύει και υπονομεύεται το διεθνές δίκαιο, οπότε θα πρέπει να δούμε το ότι αυτό επικράτησε στην Ουκρανία. Η μη διάδοση και ο αφοπλισμός ε, απειλείται για τα πυρηνικά όπλα, αλλά και τα εμπάργκο στη Λιβύη και αλλού. Power politics τι σημαίνει τεχνολογία, εμπόριο και χρηματοοικονομικά χρησιμοποιούνται ως εργαλεία διεθνού ανταγωνισμού. Πολιτικά όπλα δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα όσον αφορά τον ε, διεθνή ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών, νέες απειλές από την Ανατολή και από την ε, Κίνα, ε, ανταγωνισμός, πέραν της ε, ευκαιρία για τα παγκόσμια ζητήματα. Είναι βάλωτα τα πράγματα στη γειτονιά μας, έχουμε δυναμισμό στην Βόρειο Αφρική και επίσης θα πρέπει να δούμε ότι απειλείται η δημοκρατία και το πολυμερές ε, σύστημα διεθνών σχέσεων. Δεν είναι αυτός ο κόσμος που ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι σίγουρο ότι έχουμε ό,τι χρειάζεται για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι προκλήσει γιατί εμεί και είμαστε περήφανοι γι' αυτό έχουμε τον καλύτερο συνδυασμό ελευθερία πολιτική, οικονομική ευημερία και κοινωνική συνοχή από όλο τον κόσμο. Έχουμε του πόρου, τη στήριξη των λαών μα και ισχυρά θεσμικά όργανα και άρα αυτά είναι η βάση για μας. Και έτσι προκύπτουν οι καθημερινέ γραμμές, που εξήγηλε η νέα πρόσωπη τη Επιτροπής που θεώρησε ότι είναι γεωπολιτική υφή αυτή η, πολιτική, αυτή Ευρωπαϊκή Ένωση και μου ζήτησε να απασχίσω για μια ισχυρότερη Ευρώπη στην παγκόσμια σκηνή. Αγαπητοί βουλευτές, πώς θα γίνει αυτό. Θα πρέπει οι εθνικέ κυριαρχίε να συνδυαστούν ε, και να αναδεθούν πιο ισχυρά τα κρατημέλη και είμαι πεπισμένο ότι εάν δεν προχωρήσουμε μαζί, τότε θα καταστεί την επαύριο στον κόσμο αδύνατη η Ευρώπη. Είναι εύκολο να το λέει κανεί, αλλά είναι δύσκολο ε, να γίνει αυτή η θυσία της εθνικής κυριαρχίας. Το έλεγε και ο Ζακ ότι θα πρέπει τα λόγια να γίνονται έργα και αυτό κάθε μέρα. Όμως έτσι με συνεργασία των κρατών μελών στο Συμβούλιο θα, πετύχουμε με διαχείριση των πολιτικών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με την ε, δημοκρατική νομιμότητα που περιβάλλεται το κοινοβούλιο αυτό και πρόκειται για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και εάν επιβεβαιωθεί ο ορισμός μου τότε θα είναι στο επίκεντρο του έργου μου ως ε, αντιπροέδρου και ως υπάτο προσώπου να ενώσω την εξωτερική πολιτική των ε, κρατών μελών με την εξωτερική δράση της Επιτροπής που Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά, αλλά θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου. Η γεωπολιτική όμως ξεκινάει εδώ από το περιβόλι μας. Και γιατί αυτό, διότι πρώτα-πρώτα για να είναι κανείς σημαντικός γεωπολιτικά θα πρέπει να είναι ενωμένος περισσότερη ενότητα όπως έχουμε τώρα. Οπότε θα πρέπει και τα μικρά και τα μεγάλα κρατημέλη να πετύχουν αυτή την ενότητα και κατά δεύτερο λόγο χρειαζόμαστε συνοχή και συνέπεια μεταξύ ιστορικών πολιτικών και εξωτερικής πολιτικής. Έχουμε τα μέσα να ανταγωνιστούμε με ε, αυτή την πολιτική της δύναμης, της ισχύω, αλλά θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν μια στρατηγική. Εμεί είμαστε μια σημαντική δύναμη. Μπορούμε να κάθοσουμε στους κανόνες του παιχνιδιού και έχουμε μια ισχυρή εμπορική πολιτική και είναι δυνατή γιατί είναι κοινή. Είμαστε πρωτοπόροι για το θεματολόγιο του 2030 όσον αφορά την βιωσιμότητα, τους σχετικούς στόχους. Ε, έχουμε τον προπολογισμό μας με τον προϋποσμό των κρατών μελών και έτσι είμαστε οικονομική παγκόσμια δύναμη και η διπλωματία μας είναι από τις πιο ισχυρές. Οπότε θα πρέπει να αναβαθμίσουμε ακόμη περισσότερο τον διεθνή μας ρόλο, αλλά και την στρατιωτική μας ικανότητα για παρεμβάσεις. Δηλαδή με δύο λόγια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μάθει τη γλώσσα της ισχύω. Πολλές φορές ότι είναι το DNA της Ένωσης ε, αυτού του είδους η πολιτική και η πολυμερής μέθος, αλλά μόνοι μας τι πολυμερία έχουμε, άρα χρειαζόμαστε και συνομιλητές, αλλά πολλές φορές όμως εγκαταλείπουν ε, τους κανόνες του Πολιτείου που ισχύουν οι εταίροι μας και άλλοι είναι επιλεκτικοί ε, και δρούν σύμφωνα με τα συμφέροντά τους. Οπότε η Ευρώπη θα πρέπει να επαναορίσει το ρόλο της ε, στην σκηνή αντιπαράθεσης Κίνας-ΥΠΑ. Αντιπαράθεσης, ανταγωνισμό, όπως θέλετε, αλλά θα πρέπει να έχουμε επομένως πολυμερείς σχέσεις βάσει κανόνων να μην μας λιώσουν αυτές οι δύο υπερδυνάμεις, είπα και εκείνα. Είμαστε και θα είμαστε σύμμαχοι των ε, είπα, ισχυροί, κοντινοί σύμμαχοι. Όμως έχουμε επιφυλάξεις θεμητές για τις μονομερείς ενέργειες που κάνουν και βλάπτουν την συνεργασία. Το σύστημα επί τη βάση κάποιων κανόνων γίνεται και μπορεί να τροποποιηθεί. Επίσης, χαιρετίζουμε τη θετική κίνηση της ε, Κίνας για Ιράν και για αλλαγή του κλίματος, αλλά θα πρέπει η Κίνα να παίξει με τους κανόνες που ισχύουν. Αμοιβαιότητα, ε, ισότητα στους ε, κανόνες του παιχνιδιού. Α, για παράδειγμα, όσον αφορά επενδύσεις, εμπόριο και συνδεσιμότητα. Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, η Ευρωπαίοι ξέρουν ότι οι μεγαλύτερε προκλήσει είναι η μετανάστευση και η αλλαγή του κλίματο. Γεωπολιτικέ προκλήσει. Γιατί δεν είναι δυνατόν να λυθούν από κάποιον μεμονωμένο. Χρειαζόμαστε ε, ουδέτερη από πλευράς άνθρακα οικονομία γιατί η αλλαγή του κλίματος αναδεί το πρόβλημα του τι αναδιανομή θα γίνει κατόπιν της βιομηχανικής επανάστασης. Μεγαλύτερη πρόκληση από τότε, από τη βιομηχανική επανάσταση είναι αυτή. Οπότε έχουμε πιέσεις μεταναστευτικές, όλα αυτά θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και στο ιστορικό και στο εξωτερικό. Γι' αυτό λέω ότι όλα αυτά είναι θέματα γεωπολιτικής. Άσυλο και μετανάστευση έχουν επίσης σημαντικές επιπτώσεις. Στη Συρία έχουμε μια ανθρωπιστική τραγωδία του 2015. Ε, από τη Συρία προέκυψαν τόσοι πολλοί τον άσυλο, οπότε επιβάλλεται να υπάρξει έλεγχος, αλλά και αυθεντική συνεργασία με τις χώρες προέλευσης, κυρίως χώρες της Αφρικής και εμείς στην Ισπανία τα ξέρουμε αυτά πολύ καλά. Στο κοντινό μέλλον θα έχουμε πάνω από ένα δις περισσότερους κατοίκους στην Αφρική. Όχι να δεις συνολικά, να δεις παραπάνω και θα, θα πρέπει αυτό να το βλέπουμε μόνο σε σχέση με την μετανάστευση. Αυτό είναι και μια ευκαιρία για να υπάρξει μια συνολική στρατηγική, για να μπορούμε την παιδεία, την ασφάλεια και τι επενδύσεις όλα αυτά να τα δούμε συνολικά την απελευθερώση της γυναίκας, τη χειροφέτησή της, την, την κινητικότητα. Άρα θα πρέπει να δούμε τη συνολική εικόνα και θα πρέπει να έχουμε έτσι μια στρατηγική. Ε, έχουμε τα μέσα προς τούτο. Κάθε φορά που έχουμε κρίση μεταναστευτική, μικρή ή μεγάλη, έχουμε προβλήματα και συζητούμε τώρα για ασφάλεια και για άμυνα. Οπότε το δικό μας πλεονέκτημα είναι ότι μπορούμε να έχουμε διαμεσολάβηση, να έχουμε διαχείριση για την εξωτερική πτυχή και για την ε, ασφάλεια και με όλα αυτά βοηθούμε στην ε, ειρήνη. Έχουμε απειλές, έχουμε ε, όλα αυτά υπονομεύουν τη δημοκρατία και ξέρουμε πόσο σοβαρές είναι αυτές οι απειλές και έτσι θα προχωρήσουμε. Η άμυνα είναι θέμα παγκοσμίας ε, ασφάλειας και πολλές φορές οι απειλές ε, προέρχονται ε, από μακριά, πολύ μακριά από τα σύνορα μας. Έχουμε όμως τα μέσα για να έχουμε καλύτερη άμυνα, καλύτερε δυνατότητε άμυνας και θα προχωρήσουμε κι άλλο και υπάρχουμε 35.000 ε, Ευρωπαίους από τα κράτη-μέλη που αναλαμβάνουν διεθνώς διάφορες αποστολές και ε, ξοδεύουμε για το στρατό μας ε, περισσότερο από, την, από το, το, το μισό του, ΑΕΠ του Βελγίου, η Κίνα και όλα αυτά όμως θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ενότητα δράση, δεν θα πρέπει να έχουμε κατάτμιση των προσπαθειών, γιατί έτσι οι δαπάνε θα πιάσουν ε, τόπο. Αν τι κάνουμε όλοι μαζί με συνεργασία, να είμαστε πιο επιχειρησιακοί, να αναπτύσσουμε δυνάμεις ε, πρώτα-πρώτα εδώ από τις γειτονικές χώρε. χώρες. Λέγαμε για τους στόχους του Ελσίνκη. Θυμάστε, από το 99 μετά τον εμφύλιο της Ιουγκοσλαβίας και είπαμε ότι θα αναπτύξουν 50-60 χιλιάδες. Τότε λέγαμε. Τι έγινε με αυτό που είχαμε υποσχεθεί, ας είμαστε ξεκάθαροι. Το ΝΑΤΟ είναι και θα παραμείνει ο αγρογωνίος λίθος της συμμαχίας και της άμυνάς μας. Αλλά για να χτίσουμε μια ευρωπαϊκή άμυνα θα πρέπει να ενισχύσουμε την Ατλαντική Συμμαχία και εάν έχουμε πιο μεγάλο ειδικό βάρος εκεί θα έχουμε πιο ισορροπημένες διατλαντικές σχέσεις. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Ας μην είμαστε ο τρίτος ε, πυλώνας αυτής της ε, τριάδας σας. Είναι η Ευρώπη ένας παράγων για πολυμερή ειρηνικό κόσμο με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και έτσι να επιδιώξουμε τους, στίχους, τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό θεωρώ ότι να μην είναι κάτι σαν κήρυγμα χειρική, να είναι αυτό που λέω τώρα σήμερα τη Δευτέρα και πέραν των όσων είπατε, θέλω όλα αυτά να τα κάνω πράξη, εάν βεβαίω μου το επιτρέψετε. Thank Σας ευχαριστούμε πολύ και επειδή εμείς τηρήσατε πιστά και το χρόνο αγόρευση. Θα ξεκινήσουμε τώρα τον πρώτο γύρο των ερωτήσεων. Σας υπενθυμίζω, ένα λεπτό ο κάθε συνάδελφος, δύο λεπτά απάντηση του υποψηφίου επιτρόπου, επερώτηση ενός λεπτού και απάντηση δευτερολογία πάλι ένα λεπτό και παρακαλώ να τηρείτε όλοι το χρόνο αγόρευση. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Αντώνιο Λόπεθ από την ομάδα του ΕΛΚ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας κύριε Μπορέλ. Α περάσουμε πράγματι από τα λόγια στα έργα. Θέλετε να επικαταστήσετε την κυρία Μογκερίνη, η οποία διχειρίστηκε ε, με καταστρεφικό τρόπο την εξωτερική πολιτική. Δεν ήταν αποφασιστική σε κομμουνιστικά αυταρχικά καθεστώτα της Λατινικής Αμερικής. Ε, ουσιαστικά έκανε έναν τουρισμό. Στη Βενεζουέλα έχουμε ανθρωπιστική καταστροφή. Οι διάλογοι ε, και οι συνομιλίε έχουν αποτύχει. Και η αποτυχία ε, στην στην ε, διαχείριση ε, υπόθεσης Γουαϊδό με την Κούβα επίσης από το 2017 δεν έχουμε καμία αλλαγή στο καθεστώς. Συνεχίζει η καταστολή των κριτικών, των αντιφρονούντων τα ίδια με τον Ντανέλ Ορτέγα. Ε, τι θα κάνετε λοιπόν ε, ε, με την επιβολή κυρώσεων στις χώρες αυτές της Λατινικής Αμερικής. Ο λαϊκισμός που πλήττει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στη Λατινική Αμερική. Το βλέπουμε και σε εθνικιστική δημαγωγία εδώ στην Ευρώπη, στην Ισπανία και ιδίω στην Καταλωνία. Ε, γνωρίζω πολύ καλά και τις θέσεις σας. Τι θα κάνετε όμως ως είπα εκπρόσωπος. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ, ε, κύριε Λόπεθ Ιστουρίθ. Ξέρετε πολύ καλά ότι συμμερίζομαι τις ανησυχίες σας και για όσα είπατε για το άλλο ημισφαίριο και για όσα είπατε για τη δική μας τη χώρα. Δεν νομίζω όμως ότι έκανε τουρισμό η κυρία Μογκερίνη στην Κούβα για παράδειγμα. Όπως ξέρετε υπάρχει συμφωνία. Υπάρχει συμφωνία με την Κούβα η οποία απαιτεί περιοδικές συναντήσεις, επισκέψεις. Αυτό έκανε η κυρία Μογκερίνη. Αυτό προβλέπεται ε, στι συμφωνίε που έχει υπογράψει με την Κούβα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τη Βενεζουέλα, ε, επίση γνωρίζω πολύ καλά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα και κάνουμε πάντα το δυνατόν ώστε να πετύχουμε να γίνουν προεδρικέ εκλογέ δημοκρατικέ, εγγυημένε, ε, να μπορέσουν οι κάτοικοι της χώρας να αποφανθούν και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε την τρομερή ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα. Πάνω από 5 εκατομμύρια άτομα έχουν εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα. Πρέπει να κάνουμε αυτό που ήδη κάνουμε ουσιαστικά, δηλαδή να ασκήσουμε πολιτικέ πιέσει και να δείξουμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να διαπραγματευτούμε και να προσπαθήσουμε να γίνουν αυτέ τι προεδρικέ εκλογέ στο στομότερο δυνατόν. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ε, είπαμε ότι από 10 Ιανουαρίου ε, πάβει η δημοκρατική νομιμοποίηση του Πρόεδρου Μαδούρο πρέπει να συνεχίσουμε να επιμένουμε στην ίδια γραμμή φυσικά και απορρίπτοντα κυρώσει που θα μπορούσαν να πλήξουν ακόμη πιο κέρια και βαριά τον ε, λαό της χώρας. Ε, ατομικές μεμονωμένες κυρώσεις, ναι. Ε, έχουμε ήδη ψηφίσει το Συμβούλιο και 25 άτομα έχουν πληγεί από αυτές τις κυρώσεις και θα συνεχίσουμε να παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις. Παρότι εγώ είμαι κατά του να επιβληθούν κυρώσεις σε ένα λαό που τόσα πολλά δεινά βιώνει δεν θεωρώ ότι είναι κάτι θετικό, ούτε και τόσο θεμητό αυτό και ε, δεν νομιμοποιούμαστε να συνεχίσουμε. Τώρα για την Ικαράγω, γιατί την για τον Τάνιλ Ορτέγα, έχω μιλήσει ε, καθότι διατέλεσε πολλών εξωτερικών για αυτά τα θέματα. Η κατάσταση, θα έλεγα, στην Ικαράγω είναι ακόμα χειρότερη από αυτήν ε, στη Βενεζουέλα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπορέλ, έχετε εσείς τώρα το λόγο κύριε Λόπεθ για τη δεύτερη ερώτησή σας. Σε ό,τι αφορά τι ατομικέ κυρώσει που είπατε, ούτε το λαό τη Κούβα ούτε τη Βενεζουέλα θέλουμε να πλήξουμε. Δεν μιλάμε για τι πάμε, μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση που είχαμε μια κοινή θέση προηγουμένω. Να πληγεί το καθεστώ ουσιαστικά και περί αυτού πρόκειται. Και αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να πράττουμε. Άκουσα αυτό που είπατε για τις ατομικές ε, κυρώσεις ε, και σωστό μου φαίνεται. Ας εργαστούμε για να γίνει πράξη. Αν μου επιτρέπετε να επιμείνω λίγο ε, στην ε, προέλαση των εθνικιστικών κινημάτων. Ξέρω ότι είστε κατά ε, σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό και εντός της χώρας και εκτός. Θα μπορούσατε να μου πείτε κάτι παραπάνω. Κύριος Μπορέλ, ένα λεπτό έχετε κύριε Μπορέλ. Ναι, βεβαίως. Όπως γνωρίζετε, τα λέω έξω από τα δόντια. Outspoken το λέμε αυτό στα αγγλικά. Και τα έχω πει ντόμπρα τα πράγματα και για αυτό το θέμα και νομίζω ότι πολύ κατηγορηματικά έχω εκφραστεί και μπορώ να σας πω ότι ο ύπατος εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα έχω το καθήκον να, να ε, μιλώ για τα εσωτερικά ζητήματα κάθε μεμονωμένης χώρας. Μια γενική εικόνα και μια γενική άποψη για το τι κάνουν τα εθνικιστικά κινήματα ανά τον κόσμο, ναι, θα μπορώ να εκφράσω. Σίγουρα υπάρχουν τοπικά αίτια, υπάρχουν και κοινωνιολογικές δυναμικές που ε, ίσως υποδαβλίζουν τέτοια κινήματα. Για την Ικαράγουα ίσως μπορώ να πω κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα ε, για, το, για τα εσωτερικά μιας χώρας της Ένωσης, ακόμη και αν αυτή η χώρα είναι δική μου. Ελπίζω αυτό να το καταλαβαίνετε. Ευχαριστώ πολύ. Λέω πρόεδρος επόμενος για την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ένα λεπτό και ο ίδιος τον Νίνο Πίτσουλα. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε, κύριε Μπορέλη, στο Κοινοβούλιο. Η Ούρσολα Φοντρελάιεν, ε, οριστή πρόεδρο τη Κομισιόν, είπε ότι θα είναι γεωπολιτική η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το είπατε κι εσεί. Δηλαδή, μια ενό πιο συνεκτική συνεπή σε ό,τι αφορά την εξωτερική τη πολιτική. Και ο ύπατο εκπρόσωπος θα πρέπει να σχετίσει εσωτερικέ και εξωτερικές πτυχέ της πολιτική τη Ένωση. Καλή αυτή η προσέγγιση. Έχουμε γεωπολιτικό ανταγωνισμό όλο και περισσότερο στον πλανήτη. Εσείς είστε υπέρ τη άποψη των σιλώτων στεγανών, όπως λέγονται. Ε, δηλαδή να συνεχίσουμε φυσικά την ευημερία, να προωθούμε και αυτό όμως θα πρέπει να το κάνουμε ε, με βάση ένα σύστημα αξιών και αρχών. Ο παραδοσιακός διαχωρισμός μεταξύ των ε, ε, διαφόρων πολιτικών, εμπόριο, ανάπτυξη, εξωτερική πολιτική, πολιτική άμυνα. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται με δεδομένο το σημερινό πλαίσιο. Ευχαριστώ κύριε Μπορέλ, δύο λεπτά έχετε απάντηση βεβαίως και θα πρέπει να τα βλέπουμε ολιστικά τα πράγματα. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής είναι ακριβώς η στεγανοποίηση αυτή, η οποία βασίζεται, αν θέλετε, και στην θεσμική δομή, ότι έχουμε το Συμβούλιο με κάποιες αρμοδιότητες, την Κομισιόν με κάποιες άλλες κτλ. Όμως... Ε, πρέπει να μπορέσουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και όλες τις δυνατότητες που έχουμε ιδίω παραδείγματο χάρη την οικονομική κυριαρχία που μα ε, προσφέρει αυτό το ενιαίο νόμισμα και να διαδραματίσουμε ένα σημαντικό ρόλο. Δεν το λέω αυτό γιατί θα σας αρέσει να το, ακούτε, να το ακούσετε, αλλά γιατί πραγματικά έχω την υποχρέωση να τηρήσω το άρθρο 36 της συνθήκης που λέει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, θα πρέπει ε, να γνωμοδοτεί και οι απόψεις του να ακούγονται για τη συνδιαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής. πώληση ΣΕΙΠΕΡ. Εσείς διαμορφώνετε την εξωτερική πολιτική της Ένωσης, ιδίως δε ε, αν μιλάτε και ακούγεστε, γίνεστε και πιο κατανοητοί. Όσο πιο πολύ μιλάτε και ακούγεστε, τόσο πιο κατανοητοί γίνεστε. Δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσω τη θετική δυναμική όπως αυτή λέγεται στην πολιτική του 10 για τη λογοδοσία. Δηλαδή θα ε, έρχομαι στο Κοινοβούλιο και, την, ε, και το Συμβούλιο και την Ειδική Επιτροπή θα ε, ενημερώνω και θα ενημερώνομαι επίσης για τα πιο λεπτά ευαίσθητα ζητήματα της πολιτικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Επίσης δεσμεύομαι να εξηγώ στους βουλευτές και όλα τα επίπεδα των διαπραγματεύσεων διεθνών συμφωνιών γιατί και αυτό το απαιτεί η συνθήκη της Ένωσης. Πέντε φορές ε, το χρόνο θα έρχομαι σε κοινέ ε, συνεδριάσεις διαβούλευσης για τον προϋπολογισμό της ε, κοινής εξωτερικής πολιτικής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Θέλω να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με τις διεθνείς συμφωνίες. Δυνάμει του άρθρου 40 της Διοργανικής Συμφωνίας για την καλύτερη νομοθεσία από το 2016. Με ευχαριστώ. Έχετε κύριε Πίτσουλα τη δυνατότητα για περώτηση. Τα τελευταία 15 χρόνια, κύριε Μπορέλ, περάσαμε από έναν δακτύλιο φίλων, όπως είχε πει ο κύριος Ρωμανοπρόντη, σε έναν δακτύλιο της φωτιάς. Θα πρέπει λοιπόν να αναζωογονήσουμε την πολιτική της διεύρυνσης και γειτονίας. Κύριε Μπορέλ, εσείς είχατε προωθήσει την κοινοβουλευτική διπλωματία με τη Eurolat και τη Euromed και διακοινοβουλευτικές συναντήσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια των Κρατών Μελών. Η ερώτησή μου λοιπόν, στο πνεύμα αυτό, ποιες είναι οι απόψεις σας για την ανάγκη ε, της περαιτέρω κοινοβουλευτικοποίησης της εξωτερικής πολιτικής μας θα φροντίσετε οι πρωτοβουλίες αυτές να συνεχίσουν να εφαρμόζονται και το Κοινοβούλιο να επιβλέπει το μέλλον της ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μπορέλ, για ένα λεπτό. Νομίζω ότι ήδη είχα αρχίσει να απαντώ την ερώτηση αυτή, πρακτικά μιλώντας δηλαδή για τη συμμετοχή των βουλευτών στην ε, διαμόρφωση της κοινή εξωτερικής πολιτικής. Και αν μου επιτρέπετε να συνοψίσω και να πω ότι εγώ ζήτησα ουσιαστικά μεταξύ άλλων να, να αυτή η Ευρωλατινοαμερικανική ε, συνέλευση και άλλες τέτοιες ε, που επιτρέπουν, ε, σε, όπως και η Ευρωμεσογειακή δηλαδή, που επιτρέπουν ε, την συνάντηση ευρωπαϊκών χωρών με λατινοαμερικανικές μεσογειακές χώρες. Επίσης ζήτησα να γίνονται κοινέ διασκέψεις ε, εθνικών κοινοβουλίων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όταν ήμουν εγώ πρόεδρος ήταν δική μου πρωτοβουλία και νομίζω ότι έχει φέρει καρπούς και ο πρόεδρος της Επιτροπής σας επίσης παρίσταται στις άτυπες συνεδριάσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και ο πρόεδρος της Επιτροπής ΔΕΒΕ, διατέλεσα κατά το παρελθόν, πρόεδρος της Επιτροπής ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης, πηγαίνει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου για τα θέματα της ανάπτυξης. Ευχαριστώ πολύ. Για την ομάδα Renew. Ε, κυρία Χίλντε Βάτμαν, σε ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε κύριε Μπορέλ. Στην επιστολή της κυρίας Φόντερ Λάιεν προ εσά αναφέρεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο στρατηγική και πιο ενωμένη για να μπορεί να εξασκήσει παγκόσμια ηγεσία. Και είπατε κι εσείς ότι πρέπει να είμαστε πιο ενωμένοι, πιο ισχυροί. Ε, τα ακούω αυτό εδώ και πολύ καιρό. Η ερώτηση μου λοιπόν είναι πάρα πολύ απλή τι σκοπεύετε να κάνετε συγκεκριμένα για να επιβάλλετε την ενότητα των κρατών μελών. Αλλά θέλω απλές απαντήσεις. Μόνο έτσι θα ανακονοποιηθούν όλες οι γιατί πολλές φορές ε, ακούμε διάφορα. Δώστε μας δύο παραδείγματα δηλαδή, για να γίνετε συγκεκριμένος. Πώς θα έχουμε περισσότερη ενότητα απέναντι στη Ρωσία, πώς θα έχουμε νέα στρατηγική για τη Ρωσία και μετά για την άμυνα και την ασφάλεια, που επίσης είναι ε, προτεραιότητα για την ε, ομάδα μας, πώς θα έχουμε περισσότερη ε, ομοφωνία ως προς αυτό. Σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό για μία απάντηση. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Ορίστε. Δύο λεπτά για απάντηση. Ναι, αν υπήρχε απάντηση δίλεπτη ε, σε αυτό το ερώτημα, θα την είχε δώσει κάποιος τόσο καιρό, τέλος πάντων. Οπότε αδύνατη αποστολή μου ε, να απαντήσω σε αυτό το κοσμικό ερώτημα. Αλλά τέλος πάντων, ε, στόχος μας είναι και η διαμεσολάβηση και η δημιουργία συνένεσης, αλλά θα πρέπει να κάνουμε προτάσεις ε, για εξομάλυνση των διαφορών που μπορεί να έχουμε μεταξύ μας. Χρειαζόμαστε ε, μια κοινή στρατηγική νοοτροπία και θεώρηση. Πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, την κοσμοθεώρησή μας. Δεν έχουμε την ίδια άποψη, αλλά αν είμαστε μαζί, είμαστε μαζί γιατί έχουμε πολλά κοινά. Αλλιώ δεν θα ήμασταν εδώ που είμαστε. Άρα ξεκινάμε ε, από τους κοινούς ε, παρονομαστές Αρκεί ένα κομπιούτερ για τεχνητή νοημοσύνη ε, ίσως, αλλά ε, για να μπορέσουμε να βρούμε εμείς τις βασικές αρχές ε, της κοσμοθεωρίας μας, για να είναι κοινή η κοσμοθεωρία, νομίζω ότι χρειάζεται κάτι πολύ περισσότερο από ένα κομπιούτερ, από έναν υπολογιστή. Ε, πρέπει να δείξουμε συνέστηση, ε, να αντιληφθούμε τι τις ανάγκες του άλλου. Η Ρωσία είναι ένα παράδειγμα. Πρέπει να διατηρηθούν οι κυρώσεις στη Ρωσία όσο δεν αλλάζει στάση η χώρα και αυτό απαιτεί ενότητα, μεγάλη ενότητα, γιατί γνωρίζετε ότι μία χώρα μόνο να καταψηφίσει την επόμενη παράταση ε, καταπίπτουν ε, οι κυρώσεις. Ένα παράδειγμα που δείχνει πόσο σημαντική είναι ομοφωνία. Αν μου επιτρέπετε. Δέκα χρόνια εκπροσωπούσα σε τρεις σχηματισμούς του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τη χώρα μου. Και πιστεύω ότι το καθήκον αυτό της επίτευξης συμφωνιών έχει μεγάλη σχέση. Πρώτον με την βούληση, την επιθυμία, αλλά ε, και τη δυνατότητα να το πετύχει κανείς. Ε, εγώ ναι, πιστεύω ότι τη διαθέτω αυτή την ικανότητα. Thank ευχαριστώ. Η κυρία Βάτμανς και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η δεύτερη ερώτηση είναι πώς θα κάνετε κάτι με τα κράτη-μέλη που δεν θέλουν να συνεργαστούν για τα εξωτερικά και την άμυνα. Είστε διατεθειμένος να αναλάβετε ρίσκα γιατί καμιά φορά πρέπει να πείσουμε τα κράτη-μέλη. Π.χ. για την Ρωσία λέτε ναι, μία ψήφο αρκεί για να σταματήσουν οι κυρώσεις, αλλά για εμένα το σύστημα σου έχει δεν είναι καλό σύστημα. Έχουμε έναν ψυχρό πόλεμο με μια γειτονική χώρα. Υπάρχει μια γενιά Ρώσων νέων με αντιευρωπαϊκά αισθήματα. Καμιά φορά πρέπει να λάβουμε ρίσκα. Πώς θα πείστε τα κράτη-μέλη που δεν είναι διατεθειμένα, ε, είστε διατεθειμένα να λάβετε τέτοια ρίσκα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υποψήφιο Επιτροπή, για ένα λεπτό. Ε, βέβαια, ρισκάρουμε να μην γίνουν ε, αποδεκτές από το Συμβούλιο οι προτάσεις και να αποτελώ μειοψηφία είναι των συναδέλφων. Ας πούμε, θα προσπαθήσω σε κάποιες περιπτώσεις να μετέλθουμε το τι προβλέπει η συνθήκη όπου υπάρχει περιθώριο να μην συμφωνούμε όλοι, μην υπάρχει ομοφωνία για κυρώσεις, για ανθρώπινα δικαιώματα, για τις αποστολές της ε, ΚΕΠΑ. Οπότε εκεί δεν απαιτείται πάντοτε η ομοφωνία γιατί έχουμε ε, τις ε, περίφημες ρήτρες γέφυρα που επιτρέπουν τη λήψη απόφαση χωρίς ομοφωνία. Ε, χρειάζεται ομοφωνία για να αλλάξει η ομοφωνία όπου προβλέπεται, αλλά δεν χρειάζεται να τροποποιηθεί η συνθήκη για όλα. Δεν είμαι ένα εξ αυτών που θεωρούν ότι η δική πλειοψηφή α, είναι η πανάκια για την εξωτερική πολιτική. Και ε, χαμογελώ ε, με νόημα όταν σκέφτομαι ότι όλα αυτά τα έχουμε ε, προχωρήσει με την ε, ομοφωνία. Ε, όχι, για πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα ειρήνης και πολέμου αποφασίζουμε με δική πλειοψηφία ή τέλο πάντων με σχετική πλειοψηφία. Πράσινη. Beauty coffer. Καλώς ήρθατε κύριε Μπορέλ. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τις παρατηρήσεις σας όπου αναφέρατε τα ανθρώπινα δικαιώματα ως βασική αρχή της Ένωσης, παρά το ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν αναφέρονται στην επιστολή σας. Πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε σε αυτό. Οπωσδήποτε θα γνωρίζετε πως κάποιες παρατηρήσεις από το παρελθόν έχουν προκαλέσει κάποιες εντυπώσεις. Θα ήθελα εάν μπορούσατε να αναφερθείτε σε αυτές. Τώρα, η ερώτησή μου για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ασία. Πόση προτεραιότητα θα αποδώσετε στην στρατηγική της συνδεσιμότητας, δεδομένου του ότι μόλις υπογράψαμε και μία συμφωνία με την Ιαπωνία. Πώς θα φροντίσετε ότι θα υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση. Σας ευχαριστώ κύριος Μπορέλ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Μπουτικόφερ. Να μου πείτε σε τι αναφέρεστε και να μπορούσα να απαντήσω. Αλλιώς πώς θα σας απαντήσω. Ευχαριστώ να σας πω. Τώρα όσον αφορά την συνδεσιμότητα. Οφείλω να σα πω ότι πρόκειται για την πιο μεγάλη τάση του 21ου αιώνα. Αυτό θα καθορίσει την δεκαετία του 2030, ε, η διασύνδεση, η συνδεσιμότητα του κόσμου, κάτι που θα μας δείξει τι ροές θα υπάρχουν, τι στάνταρ θα υπάρχουν για παγκόσμια διακυβέρνηση και έχουμε διακυβέρνηση σχετικά. EU Connecting Europe λέγεται, σε συνεργασία με Ασία, τον Οκτώβριο του 2018. Διόλα γιατί Πού βασίζεται, ποιοι είναι βιωσιμότητα, νοητή και τήρηση κάποιων κανόνων. Τι θα πει βιωσιμότητα, βιωσιμότητα από πάσα απόψεως ε, δημιουργικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ε, συνολικά. Δεν είναι μόνο λιμάνια και γέφυρες και υποδομές, αυτά που λέγαμε μια φορά και ένα καιρό. Όχι, το λέμε για δίκτυα ψηφιακής εποχής και σύνδεση του ανθρώπου με τον άνθρωπο. Επίσης, τι εννοούμε με πλέγμα κανόνων, να υπάρχει ένα τέτοιο πλαίσιο, τόσο ώστε να μπορεί ο κόσμος να έχει κάποια ελευθερία, αλλά και οι εταιρείε που θέλουν να επενδύσουν ε, μέσα σε κλίμα ασφάλειας. Επίσης, ε, θα πρέπει να κάνουμε και άλλα βήματα προόδου με τρεις ε, συγκεκριμένου αξονες άξονες. Πρώτα-πρώτα, να χτίσουμε κάποια δίκτυα με την Ασία το πεδίο της ενέργειας, της ψηφιοποίησης και των ε, διανθρωπίνων σχέσεων. Επίσης, να συνεργαστούμε στενά με τους ε, εταίρους μας. Αναφέρατε την Ιαπωνία, αυτό έγινε πραγματικισμένο μας, 27 Ιανουαρίου, να κάνουμε το ίδιο με Ινδία, Κορέα και τις χώρες ΑΣΕΑΝ. Κατά τρίτο λόγο. Thank you λήξη χρόνου. Επόμενη ερώτηση. Κύριε έρχεται η ερώτηση. Είμαι σίγουρος, κύριε Μπορέλ, πως και το τρίτο σημείο θα το αναφέρετε στην δεύτερη απάντηση. Και αν ε, με ρωτούσατε το τι πρόσεξα εγώ, πρόσεξα αυτό που είπατε για τους τέσσερις νεκρούς Ινδούς. Αλλά να επανέλθω έχει ασκηθεί κριτική στις ε, μεμονωμένες ε, πολιτικές ε, από τους συναδέλφους μου και το είπατε και εσείς. Όμως αυτό το οποίο βλέπω εδώ πέρα το οποίο δεν υπήρχε πριν από πέντε χρόνια της κυρίας Μογκερίνη είναι το εξή ότι ως αντιπρόεδρος θα καθοδηγείτε όλες τις πολιτικές που αφορούν τις εξωτερικές σχέσεις. Αυτό υπήρχε στην αποστολή της κυρίας Μογκερίνη, αλλά όχι στην δική σας. Θα μπορείτε εσείς να καθοδηγείτε την εξωτερική πολιτική για να μην έχουμε μεμονωμένη άσκηση πολιτικής ανακλάδου. Σας ευχαριστώ κύριος Μπορέλ για ένα λεπτό. Το άρθρο 18 της συνθήκης δεν χρειάζεται κάποιο είδου ε, επιστολή ανάθεσης ε, της αποστολής ε, εκεί ορίζεται ότι εγώ έχω την αρμοδιότητα του συντονισμού της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα πράγμα είναι οι εξωτερικές πολιτικές και άλλο ιστορικές πολιτικές που έχουν εξωτερική διάσταση. Ε, βέβαια, για τις τελευταίες θα πρέπει να συνεργαστώ με την Πρόεδρο. Επίσης η επαρκής χρηματοδότηση δεν θα πρέπει το θέμα αυτό να το παραμελούμε. Τώρα στην Κροατία κατασκευάζεται μια μεγάλη ε, γέφυρα 800 ε, εκατομμυρίων. Τα 400 ε, κάνουμε συνεργαζόμαστε με Κινέζους ε, και οι εργαζόμενοι, οι Κινέζοι μένουν σε ένα πλοίο που είναι δεμένο εκεί στο εργοτάξιο. Βέβαια δεν ξεχνούμε τι έγινε με τον Ινδό και είπαμε ότι εμείς δεν θα γίνουμε ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης Άλλωστε υπάρχει προστορία αντιπαραθέσεων. Ευχαριστώ. Από την ομάδα ID, ο κύριος Μαριάννη. Ευχαριστώ. Πέρυσι το Μάιο, κύριε Μπορέλ, στον Ισπανικό τύπο περιγράφατε τη Ρωσία σε μια συνέντευξή σας ω τον παλαιό μας εχθρό. Υπάρχει ένας πραγματικός εχθρός, αν με επιτρέπετε, που ποτέ δεν έχει κατονομαστεί ε, σε αυτά τα 45 λεπτά μέχρι τώρα, που είναι η ριζοσπαστική Ισλαμική τρομοκρατία στη Γαλλία. Ε, χτύπησαν πάλι τις τελευταίες μέρες, όπως και σε όλες τις χώρες μας. Είναι σήμερα μια πραγματική απειλή. Πενθυμίζω ότι η έκθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιουλίου λέει ότι στους τελευταίους Συριακούς θύλακες Έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό ε, τρομοκρατών μαχητών, ξένων μαχητών στον κόσμο. Ποιος είναι λοιπόν για σας ο χειρότερος εχθρός, ε, η Ρωσία ή η τρομοκρατία. Και αν είναι τρομοκρατία, τι θα κάνετε για να επηρεάσετε χώρε που τον έχουν χρηματοδοτήσει ή τον χρηματοδοτούν αυτόν τον εχθρό, όπω η Σαουδική Αραβία, ε, το Κατάρ ή η Τουρκία, που έχει έναν αμφίβολο, αμφίσιμο ρόλο. Δύο λεπτά έχετε, κύριε Μπορέ. Ακούστε. Δεν είπα ποτέ εγώ ότι ήταν εχθρός ε, της χώρας μου τουλάχιστον ε, η Ρωσία, για την Ευρώπη μίλαγα και το ίδιο λέω και ε, εδώ ενώπιόν σας. Οι Ηνωμένε Πολιτείε τώρα έχουν μία κάπως πιο ασαφή θέση σε σχέση με το παρελθόν. Υπάρχουν νέες απλές που αναδύονται από την Ανατολή κτλ. Και χρειάστηκε να δώσει εξηγήσει ε, ο πρέσβης. Εγώ δεν είπα ε, ότι είναι η Ρωσία εχθρός ε, της Ισπανίας, αλλά ισχύει ότι υπάρχουν νέες απειλές, γιατί αν δεν υπάρχουν αυτές οι νέες απειλές, τότε τι κάνουν τα μαχητικά μας F-18 και τα Λέοπαρτ του Ισπανικού στρατού στην Εστονία και στη Λιθουανία, για να πιούν καφεδάκι πήγαν εκεί ή πήγανε γιατί υπάρχει απειλή και η Ατλαντική Συμμαχία έχει να την αντιμετωπίσει και θέλει ε, τη ε, συνοδρομή Καναδών και Ισπανών ή την έχει εξασφαλίσει ε, πραγματικά ε, και δεν νιώθουν το ίδιο ίσως οι με τους Ισπανούς αλλά είναι σημαντικό ότι αυτά τα Ισπανικά στρατεύματα συμμετέχουν ε, στην αντιμετώπιση αυτού που για πολλούς Ευρωπαίους είναι απειλή, θεωρείται ως απειλή. Και νομίζω ότι περέβαλαν ε, όταν ε, κάλεσαν τον πρέσβη οι Ρώσοι για να δικαιολογήσει αυτά τα οποία υπόθηκαν. Το θέμα είναι ότι εμείς βλέπουμε πιο ε, κοντά ίσως και το νιώθουμε περισσότερο ε, τις ε, περιπόλους και όλους αυτούς τους στρατιώτες περιπολούν γιατί φοβούνται την τρομοκρατία και σίγουρα είναι κάτι που το ζούμε πιο κοντά. Ε, θα πρέπει να έχουμε σίγουρα ε, συνεργασία με αυτές τις χώρες κατά το παρελθόν ίσως φιλοξένησαν αυτούς τους ε, μαχητές και πρέπει να υπάρχει συνεννόηση. Δυστυχώς διακόπτεται. Κύριε Μαριανή, Άρα τρομοκρατία είναι ο βασικό εχθρό, αν συνάγω σωστά. Επομένω, αν γίνεται, είπα το εκπρόσωπο, επανέρχομαι στο ερώτημα, τι θα κάνετε με χώρε όπω είναι η Σαουδική Αραβία, Κατάρι, ίσω και η Τουρκία που έχουν μια αμφιβολή θέση. Σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση τη τρομοκρατία, είναι ένα θέμα το οποίο η Ευρώπη θα πρέπει να επενδύσει. Έχει βαρύνουσα θέση, αλλά δεν επηρεάζει τόσο πολύ τα πράγματα. Ε, είναι ανεπαρκής για να μην πω ανύπαρκτη ε, η δική μας δράση σε ό,τι αφορά αυτές τις τρίτες χώρες ε, και τι γίνεται με αυτούς τους ε, υπηκόους των χωρών της Ένωσης που είναι σε αυτές τις χώρες που υποθάρουν την τρομοκρατία. Πρέπει να τους αφήσουμε εκεί να τους επαναπατρίσουμε. Τι λέτε. Απάντηση. Ακούστε, στο πρώτο ερώτημα εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι ασαφής η αμφιβολή θέση της Τουρκίας ό,τι αφορά την τρομοκρατία. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπήρξαν διαδικασίες δραστηριότητας, ε, η χρηματοδότηση που ευνόησαν τελικά ίσως το πρόσφορο έδαφος ε, αυτό από το οποίο βγαίνουν ε, οι νέοι αυτοί τρομοκράτες, αλλά θα πρέπει να ε, αγωνιστούμε από κοινό κατά του κοινού εχθρού. Ισλαμιστές, τρομοκράτες, πολύ πιο πολλούς μουσουλμάνους από ότι χριστιανούς έχουν δολοφονήσει, δηλαδή πολύ περισσότερα θύματα της τρομοκρατίας στην Αφρική, στην Ανατολική Αφρική κτλ. Δεν είναι Ευρωπαίοι. Πρέπει να δούμε τα νούμερα και το άλλο ερώτημά σας μπορείτε να το επαναλάβετε. Α, ναι. Ναι, έχουμε κάποιου εμεί, αρκετού ε, στην Ισπανία, θα του επαναπατρίσουμε. Γιατί κάθε Ισπανό υπήκο είναι Ισπανό υπήκο και πρέπει να ε, προστατευθεί. Και αν έχει λογαριασμού με τη δικαιοσύνη, θα πρέπει πράγματι να εξασφαλίσουμε ότι θα δικαστεί. Ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο για το ECR στην κυρία Φωτίνκα. Thank you, σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, εδώ πέρα θέλουμε να ακολουθούμε τις ρήτρες του ΟΗΕ. Έχουμε την στρατηγική ναυτικής ασφαλείας και πολλές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στην θάλασσα, στην νότια συνική θάλασσα Έχουμε ναι, έχουμε μπλοκάρισμα των στενών της Αζωφικής, ε, ναι, στον ναι. κόλπο του Άντεν ε, και αλλού, αλλά και στον Βιστούλα, εκεί στη Λιμνοθάλασσα τα ίδια συμβαίνουν. Πώς ε, θα προστατεύσετε τα ναυτικά συμφέροντα της Ένωσης παγκοσμίως Νομίζω η εξωτερική πτυχή της θαλάσσιας στρατηγικής μας είναι άμεση δική σας ευθύνη. Σας ευχαριστώ κύριε Μπορέλ. Δύο λεπτά. Ε, ευχαριστώ. Ναι. Να προστατεύσουμε αυτές τις κινήσεις σε κάθε ήπειρο και σε όλες τις θάλασσες είναι Ηράκλειος άθλος. Χρειάζεται τεράστια ε, δυνατότητα στη Έχουμε βέβαια την ε, επιχείρηση ε, Αταλάντη κατά των πειρατών στο κύριο της Αφρικής και έχουμε σκάφη ισπανικά τα οποία επιτελούν σημαντικό έργο όσον αφορά το τι γίνεται σε εκείνη τη γωνία του κόσμου. Δεν μπορούμε να αναπτύξουμε στόλους εκεί, αλλά σας σας ανησυχεί το ορμούς Εκεί υπάρχει ο Αμερικανικός στόλος προστασίας. Εμείς δεν συμμετέχουμε σε αυτή την επιχείρηση. Εις δε το Συμβούλιο προσφάτως συζητήσαμε το πώς θα υπάρξει και η Ευρωπαϊκή Ναυτική Δύναμη εκεί. Δεν επιτεύχθηκε όμως ε, συμφωνία και Ούτε νομίζω, τουλάχιστον στο άμεσο δεν θα υπάρξει συμφωνία. Τι μπορούμε να κάνουμε. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να συγκαλέσουμε μια διάσκεψη περιφερειακή, ε, να συμμετάσχουμε και όλα τα μέρη να αρχίσουν έναν διάλογο με στόχο την αποκλιμάκωση, το να στείλουμε και εμείς εκεί ναυτικές δυνάμεις ε, τι θα γίνει, τι να έχουμε, την ε, σπίθα που θα, που θα φέρει την έκρηξη στην πρωταποθήκη, καλύτερα να προσπαθήσουμε να έχουμε αποκλιμάκωση, μήπως και τα βρουν τα αντιπαρατηθέμενα μέρη. Ούτως ώστε να έχουμε μια ευρύτερη γεωπολιτική ισορροπία. Μπορούμε εκεί να παίξουμε αυτόν τον σημαντικό ρόλο. Λέει ο κύριος Μπορέλ, φωτίγκα. Έχει επερώτηση. Ε, ευχαριστώ. Πάλι η Ρωσία μπλοκάρει την ελευθερία της συναυσιπλοείας στην Αζωφική και στον Βιστούλα. Τι άποψη έχετε για τις κυρώσεις κατά της ε, Ρωσίας λόγω της ε, στάσης της απέναντι στην Ουκρανία. Κύριε Μπορέλ. Δεν αναφέρθηκα σε αυτή τη γωνία του κόσμου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό μέρος για την Ευρώπη. Όσον αφορά τις κυρώσεις της Ρωσίας, το προείπα και δεν ε, με δυσκολεύει το ξαναπώ. Θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε σχέση με την διατήρηση αυτών των κυρώσεων που ξεκίνησαν πρώτα-πρώτα για την παραμή προσάρτηση της Κρυμαίας και διότι παρεβιάστη η εθνική κυριαρχία της Ουκρανίας. Εάν δεν η Ρωσία, τότε θα πρέπει να συνεχίσουν να ισχύσουν αυτές οι κυρώσεις. Και δεν χρειάζεται η ομοφωνία πολιτική Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε τις πέντε αρχές της σχέσης μας με τη Ρωσία. Δεν έχουμε ένα πράγμα με έναν άξονα. Και επίσης ε, λέμε ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε μαζί με τη Ρωσία σε όλα τα μέτωπα που υπάρχει περιθώριο διαλόγου. Σας ευχαριστώ. Να δώσω τον λόγο τώρα στην κυρία Βιγενοέβα Ρουής από την ΚΟΕ. Τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες αυτής της κούρσας εξοπλισμών. Η ΕΠΑ και η Ρωσία παραβιάζουν τις ε, συμφωνίες μη διάδοσης των πυρηνικών επίσης πολλαπλασιάζονται οι πολεμικές αναμετρήσεις με πολλές μορφές σε πολλά μέρη. Όλο ένα και περισσότερο ασταθής γίνεται η υδρόγειος. Έχουμε επίσης το φοβερό ότι ο Τραμπ τώρα κάνει πλάτες στην Τουρκία ούτως ώστε αυτή να επιτεθεί στους Κούρδους στη Βόρεια Συρία. Εσείς τι λέτε, δεν πρέπει εμείς να γίνουμε ένα φρένο ή τέλος πάντων να γίνουμε πηγή παγκόσμιας ασφάλειας για έλεγχο εξοπλισμών και για την ε, Τουρκία. Δεν θα πρέπει αυτή η επικείμενη επίθεση να καταδικαστεί και να παγώσουμε τον, ε, τη χρηματοδότησή της. Έχετε δίκιο, κυρία βουλευτή. Όντως, μπαίνουμε σε φάση πυρηνικής αστάθειας και είναι πολύ βαριές αυτές τις κουβέντες, αλλά ισχύει αυτό. Οι συμφωνίες, η μία μετά την άλλη, οι συμφωνίες που είχαν ένα δίκτυο πρόληψης για την αύξηση εξοπλισμών και λοιπά και για τη χρήση καταπίπτουν η μία μετά την άλλη οπότε. Γι' αυτό σας λέω. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσουμε να διαδραματίσουμε αυτόν τον ρόλο του πώς η Συμφωνία Μη Διάδοσης των Πυρηνικών να παρεκταθεί. Αφοπλισμός, η ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας και μη διάδοση. αυτή οι τρεις πυλώνες της συμφωνίας. Ε, και θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με το Ιράν, πώς θα ε, συνεχιστεί να ισχύει η συμφωνία, να συνεχίζουμε να πασχίζουμε ούτως ώστε να τεθεί σε ισχύει η σχετική συμφωνία για τις πυρηνικές δοκιμές. Πάντως ξέρετε ότι δεν υπάρχει κοινή θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη συμφωνία απαγόρευση των πυρηνικών, οπότε δεν έχουμε κοινή θέση. Μόνο μία ευρωπαϊκή χώρα προωθεί την σύναψη δύο συμφωνίας. Οι υπόλοιποι όχι. Έτσι είναι τα πράγματα στο Συμβούλιο. Ε, γι' αυτό σας λέω, δύσκολα θα αλλάξει η κατάσταση. Φυσικά και είμαι κατά των πυρηνικών και φανταρώ και οι περισσότεροι εξημών. Αλλά αυτό ισχύει στο Συμβουλίο. Τώρα για την Τουρκία. Ιράκ, Τουρκία. Είπα σήμερα το πρωί το έμαθα. Η κατάσταση είναι εξόχως σοβαρή. Έδωσε το πράσινο φως η Αμερική για να μπουν οι Τούρκοι στο Ιράκ. Ακόμα ένα περιστατικό επομένως για το οποίο θα πρέπει να δει η Ευρώπη τι θα κάνει να λύσει το πρόβλημα. Ο πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση. Ευχαριστώ. Η επερώτηση. Ότι τη σήμερα ημέρα χρειαζόμαστε παράξει περισσότερο από πότε εσείς ήσασταν στη χώρα μας υπουργό και δώσα το πράσινο φως για πώληση όπλων ισπανικών στη Σαουδική Αραβία που ξέρουμε ότι είχαμε ε, από τη χρήση των οπλαυτών πάνω από 200.000 νεκρούς και κατα, καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εσείς τι λέτε. Έχουμε τη συμφωνία του Δεκεμβρίου του 8 όσον αφορά κοινού κανόνες για την εξαγωγή όπλων. Και θεωρούμε ότι η Ισπανία ακόμα δεν έχει προσυπογράψει ενώ το έχει υποσχεθεί τη συμφωνία για τα πυρηνικά. Σήμερα δε όσον αφορά τη συμφωνία της μη διάδοσης χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα. Τώρα δεν νομίζετε ότι έχουμε περισσότερες δυνατότητε για να το κάνουμε αυτό. Σας ευχαριστώ. Όπως και εσείς και εγώ το γνωρίζω ότι έτσι είναι τα πράγματα, αλλά δεν είναι η θέση μου τώρα να σας εξηγήσω την ισπανική εξωτερική πολιτική. Πάντως, η δική μου κυβέρνηση δεν πώλησε άλλα όπλα. Απλώς ίσχυσαν τα όσα είχε συμφωνήσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Θέλει η κυβέρνηση να προσυμπορεύσει τη συμφωνία, και να δούμε αν θα συνεχιστεί η συμφωνία, γιατί είχε γίνει μια συνάντηση προς τούτο πολύ σημαντικό. Άρα, εμείς θέλουμε να συνεχιστεί ότι ισχύει. Όσον αφορά τώρα την εξαγωγή των όπλων, Νομίζω ότι θα πρέπει όχι μόνο να συνεχίσει να ισχύει η συμφωνία του 8, αλλά θα πρέπει να την επικαιροποιήσουμε γιατί το 8 είναι μακριά, άρα χρειάζεται ένα κοινό πλαίσιο ευρωπαϊκό για τι εξαγωγέ και άρα θα πρέπει να αναθεωρηθεί η συμφωνία του 8. Σας ευχαριστώ κύριε υποψήφια επίτροπε. Περνάμε τώρα στον δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην κυρία Καλνιέτε για το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαι κύριε Μπορέλ, εδώ. Τα Δυτικά Βαλκάνια είναι μια περιοχή προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της προοπτικής ένταξης. Στην προηγούμενη θέση σας ως Υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας εκπροσωπήσατε μια χώρα η οποία δεν αναγνώριζε το κοσφοπόεδιο. Ως ε, ύπατος εκπρόσωπος ε, θεωρείτε ότι θα μπορέσετε να πείστε την κυβέρνηση της Ισπανίας να αναγνωρίσει το κοσφοπέδιο εάν συνεχίσει η μη αναγνώριση από την Ισπανία αναπόφευκτα η δική σας η αξιοπιστία και η ακαιρεότητα της πολιτικής σας θα αμφισβητηθεί. Ποια λύση προτείνετε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπορέλ για δύο λεπτά. Η αναγνώριση του κοσφοπεδίου είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Γνωρίζετε ότι διαφέρουμε στην αναγνώριση, αλλά είμαστε ενωμένοι στις επαφές. Και βεβαίω σαφέ είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία με την Σερβία. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την προτεραιότητα. Μάλιστα η πρώτη μου επίσκεψη θα είναι στην Πριστίνα. Γνωρίζω τη Σερβία πάρα πολύ καλά. Είχα καλέσει τον Πρωθυπουργό της χώρας να πάει σε ένα Ισπανικό Πανεπιστήμιο. Δεν έχω πάει ποτέ στο Κοσμοπέδιο για προφανείς λόγους, αλλά θα είναι η πρώτη μου επίσκεψη γιατί θεωρώ ότι εμείς ως Ευρωπαίοι αν δεν μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα με στην γειτονιά μας, δύσκολα θα μπορέσουμε να είμαστε μια γεωπολιτική δύναμη. Τελικά σημασία δεν έχει το τι κάνει η Ισπανία, γιατί όσον αφορά την... Ε, όσο η Κίνα, η Ρωσία και η Ινδία δεν το αναγνωρίζουν, δεν θα είναι κράτος. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε σκληρά για να συνεχίσουμε τις συνομιλίες το κοσφοπέδιο πρέπει ακριβώς να αναγνωρίσει τα καθήκοντά του και να περάσει σε έναν ειλικρινή διάλογο ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια και κρατάει εδώ και πάρα πολύ καιρό για να είστε σίγουρος ότι αυτό θα είναι ένα από τα ζητήματα που θα με απασχολήσει πάρα πολύ γιατί το τωρινό καθεστώ δεν μπορεί να συνεχίσει και χαίρομαι ιδιαίτερος για το ότι χτες το κοσφοπέδιο ε, διεξήγαγε δημοκρατικές εκλογές. Πρέπει να συμφωνήσουμε με την Σερβία και το Κοσμοπέδιο. Σας ευχαριστώ κυρία Καλνιέτη, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Μπορέλα. Αναφέρατε Κίνα, Ρωσία και λοιπές που επίσης δεν αναγνωρίζουν το κοσφοπέδιο, αλλά αυτές δεν είναι κράτη-μέλη. Εγώ είμαι πρώην διπλωμάτης και θα προτιμούσα να σας ρωτώ για τις ε, προκλήσεις εξωτερικής πολιτικής. Όμως ε, πρέπει να θέσω ένα θέμα ακαιρεότητας. Τι συμπεράσματα έχετε βγάλει από την υπόθεση της Ισπανίας ε, για την κατάχρηση εμπιστευτικών εταιρικών πληροφοριών. Στο αξίωμά σας θα έχετε πολύ πιο σημαντικές πληροφορίες στην διάθεσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ πάντοτε αρνήθηκα κάτι τέτοιο. Ξέρω ότι μου επευλήθη κύρωση από αυτού, αλλά μιλάμε για μια συναλλαγή 9.000 ευρώ που το 90, μάλλον ήταν το 7% του χαρτοφυλακίου μου. και το 93% το, διατέλεσα, το διατήρησα συγγνώμη, μέχρι που έχασε την ε, αξία του. Και θα το δει και στι φορολογικέ μου δηλώσει. Έχασα 300.000 ευρώ. Κάποιο που έχει τέτοιε προνομιακέ πληροφορίε στα χέρια του, τι πιστεύετε, χρησιμοποιεί για να απολύσει μόνο το 7% του χαρτοφυλακίου του και να χάσει το 93% των υπόλοιπων για μια συναλλαγή 9.000 ευρώ που δεν έγινε σε μια σωστή χρονική στιγμή σίγουρα, αλλά όταν χάνεις ταυτόχρονα το 93%. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται σε τόσο πολύ εμπιστευτικές πληροφορίες που δεν ήταν και καν δικό μου, ήταν ε, η επιτέως σύζυγός μου που δεν διαχειριζόταν. Μακάρι να είχαμε τέτοιου είδου προνομικέ πληροφορίες στα χέρια μα. γιατί και αυτή έχασε 80% του χαρτοφυλακίου. Ευχαριστώ πολύ. Σας και... Ευχαριστώ. Δίνω τον λόγο τώρα στην κυρία Μαρία Αρένα, πρόεδρο της Υποεπιτροπής Ανδρομικών Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπορέλ. Είπατε δεν κάνετε κήρυγμα τη Κυριακή και δεν με ενδιαφέρει κιόλα αυτό. Γι' αυτό με ενδιαφέρει αυτό που λέτε σήμερα Δευτέρα. Και ιδίω σε, σε ό,τι αφορά τη δική για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και για το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων που γίνεται λόγο σε σεβασμό στα ανθρωπίνα δικαιώματα και στι αρχέ τη δημοκρατία, τη ισότητα, ε, του κράτου δικαίου, ε, που είναι οι κατευθυντήριε ε, αξίε και αρχέ ε, και καθοδηγούν τι δράσει μα εντό και εκτό συνόρων. Το άρθρο 21 τη Συνθήκη Ευρωπαϊκή Ένωση, επίση μιλά για την πράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πρέπει να είναι στο επίκεντρο του διαλόγου και των σχέσεών μα με τρίτε χώρε, είτε σε ό,τι αφορά διαπραγματεύσεις για εμπορικές, οικονομικές συμφωνίες ή είτε για συζητήσεις για τη μεταναστευτική πολιτική. Άρα, ερώτημα, τι μέτρα θα λάβετε ώστε το σύνολο ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά το σύνολο να σέβεται αυτές ε, τις διατάξεις και οι πολιτικές άλλων επιτρόπων ε, και ιδίως του αρμοδίου για το Εθνές Εμπόριο Επιτρόπου να μην παραβιάζουν τις αρχές αυτές, δηλαδή τις αρχές που άπτονται του ασμούς στα ανθρώπινα δικαιώματα. Απάντηση. Ναι, καταλαβαίνω, κυρία Βουλευτά. Καταλαβαίνω ε, την ε, επιφυλακτικότητά σας ε, γιατί έχουμε από τη μια την άτεκτη πραγματικότητα και τις αναπλατρήτες αρχές και πρέπει να βρούμε πάντοτε την ισορροπία μεταξύ αυτών. Αλλά νομίζω το πρώτο που πρέπει να έχουμε είναι αρχές. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα είναι ένας φάρος, σύμβολο προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρωτοστατή και αυτό πρέπει να το καταστήσουμε αναπόσπαστο τμήμα όλων των ε, πολιτικών που εφαρμόζουμε. Προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, δεν ε, ε, προασπίζουμε σε κάποια γωνιέ του πλανήτη. Είναι στο επίκεντρο όλων των πολιτικών. Και νομίζω ότι πρέπει να δρομολογηθεί ένα νέο σχέδιο δράση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ζητήσω τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και τη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε διμερείς συμφωνίες έχουμε διατάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχουμε χώρες ε, που δικαιούνται ε, προνομιακή μεταχείρισης. Πρέπει να σέβονται ε, τις διατάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το εργασιακό δίκαιο. Θα μου πείτε ναι, αυτά όλα είναι γραπτά αλλά δεν εφαρμόζονται. Ναι, αλλά αυτοί που δεν τηρούν τις διατάξεις θα πρέπει να έχουν υπόψη τους και τις επιπτώσεις. Σας διαβεβαιώ, για μένα τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι το επιστέγασμα απλά μια εμπορική συμφωνία, οικονομική συμφωνία, αλλά είναι αναπόσπαστο τμήμα, όχι μόνο κατά τη σύνταξη συμφωνία, αλλά και κατά την παρακολούθηση τη εφαρμογή τη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πράγματι πρωτοστάτησε ε, στις προσπάθειες αυτές, παραδείγματος χάρη, κατά της παιδικής εργασίας και για την προστασία των κοινωνικών ε, περιβαλλοντικών ε, διατάξεων. Αυτό είναι κάτι που προσλαμβάνει όλο και μεγαλύτερη σημασία, διότι ενίοτε ακριβώς επί τη βάση της παραβίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, παίζεται και η ανταγωνιστικότητα. Όταν παραβιάζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί να έχουν περισσότερο κέρδος ενδεχομένω. Αυτό λοιπόν ε, έχει να κάνει και με το γεωπολιτικό παιχνίδι όπως παίζεται σήμερα. Ευχαριστώ. Συμπληρωματική ερώτηση. Ναι, ευχαριστώ. Σύντομα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κληθεί να συζητήσει με χώρες όπως Ινδία, Βραζιλία, Κίνα, Ισραήλ, Καζακστάν, Ρωσία, λίγες μόνο αναφέρω, στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. Με τις χώρες αυτές έχουμε συνάψει συμφωνίες που περιλαμβάνουν ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο σεβασμό του ω ένα σημαντικό κομμάτι των συμφωνιών. Συγκεκριμένα, πώ θα φροντίσουν να εφαρμόζονται οι ρήτρε αυτέ που μέχρι τώρα δεν έτυχαν καμία παρακολούθηση στο πλαίσιο εφαρμογή των συμφωνιών αυτών για να είναι αξιόπιστη ένωση σε αυτό το θέμα. Τι θα κάνετε Πώ θα αναφέρεστε στι διμερείς επαφέ που θα έχετε με αυτέ τι χώρε ακριβώ στη ρήτρα για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, Παρά τους φόβους ε, που τυχόν έχετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται αντιληπτή ως ε, ένας αξιόπιστος εταίρος από πρασπίσεις ανθρώπινα δικαιώματα. Μπορεί και να μην κάνουμε πάρα πολλά, ευτυχώς όμως που είμαστε εκεί και κάτι κάνουμε. Εμείς. Μου είπατε συγκεκριμένα τι θα κάνω. Αυτό που θα κάνω λοιπόν είναι η ρήτρα αυτή για τα ανθρώπινα δικαιώματα να συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις διμερείς εμπορικές συμφωνίες και ο διάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με τις πολιτικές κοινωνικο-οικονομικές ε, σχέσεις με τις χώρες αυτές να οδηγηθεί σε ένα ε, αποτέλεσμα που θα λαμβάνει υπόψη και τις ιδιαιτερότητες της κάθε Έχουμε ένα σχέδιο δράσης για την περίοδο από το 2020 το 2024. Έχουμε πολλά σχέδια δράσης ε, βέβαια, αλλά αυτά θα πρέπει να τα δούμε στην πράξη. Πώς μεταφράζονται. Και καλό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζητώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεργαστεί, να εργαστεί μαζί μου, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά να είναι φάρος της προστασίας των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων στον κόσμο. Thank Σας ευχαριστώ. Τώρα δίνω τον λόγο στην κυρία Ναταλή Λουαζό, μέλος της ομάδας Ρινιού και ε, της ε, Υποεπιτροπής Άμυνας και Ασφαλείας. Ευχαριστώ Πρόεδρε κύριε Μπορέλ. Κύριε Φοντερ Λάιεν, ξεκάθαρα είπε ότι έχει την φιλοδοξία να είναι επικεφαλή μιας γεωπολιτικής επιτροπής από πλευρά ασφαλεία και άμυνα αυτό που θα πρέπει περισσότερο να συνειδητοποιήσουμε στην Ευρώπη για να αναβαθμίσουμε την κοινή άμυνα σήμερα είναι ε, κάτι που συμφωνούμε όλοι. Το 2016 είπαμε ότι έτσι θα πρέπει να έχουμε ως στόχο την στρατηγική αυτονομία και έτσι ε, χαράξαμε κάποια μέσα πολιτικής ε, την μόνιμη συνεργασία, το, Ταμείο Άμυνας, οπότε οφείλουμε τώρα να ενεργήσουμε τη βάση αυτών των μέσων που στη διάθεσή μας, αλλά σήμερα αυτό το οποίο δεν ισχύει, δεν υπάρχει μια νοοτροπία κοινή στρατηγική, ένα κοινό δόγμα. Επανειλημμένα το κοινοβούλιο είπε στην ε, υπάτη εκπρόσωπο κάτι να κάνει σε σχέση με ένα, μια λευκή βίβλο για την Εσείς πρόκειται να βοηθήσετε τόσο ώστε να υπάρξει αυτή η λευκή βίβλος. Κύρια Βουλευτά, όντως δεν έχουμε, δεν έχουμε αυτήν την κοινή στρατηγική νοοτροπία. Και έχουμε ένα πρόγραμμα αμυντικό, έχουμε επιχειρησιακό, έχουμε τις ε, ε, αποστολές μας για ασφάλεια και άμυνα ε, και θα πρέπει να κάνουμε βήματα πρόοδου οπότε. Ο κύριος Λουλαμή είπε τις πρόλες, θα πρέπει να προχωρήσουμε να μην κοινοτικοποιήσουμε το διακυβερνητικό. Ούτε το αντίστροφο. Ούτε το αντίστροφο να αφήσουμε ότι είναι διακυβερνητικό, διακυβερνητικό. Επομένως, γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να βρούμε μία πλατφόρμα, τα στρατηγικά μας προγράμματα και να δούμε αν αυτά αρκούν ή αν θα πρέπει να κάνουμε και άλλα βήματα. Κατά τη γνώμη μου, έχει αποδειχθεί σε εθνικό επίπεδο ότι αξίζει μια λευκή βίβλος. Είναι μία μέθοδος που θα μπορούσε να επηρεάσει το τι θα κάνουμε στο μέλλον. Όμως γνωρίζετε πολύ καλά ότι πρόκειται για κάτι δύσκολο. Και θα πρέπει πριν ξεκινήσουμε τέτοιο εγχείρημα να δούμε κατά πόσο υπάρχουν τα απαραίτητα από πλευρά στρατιωτικής, διοικητικής, πολιτικής. Οπότε, το θέμα είναι κατά πόσο να κρατήμεται είναι αποφασισμένα. Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, εάν δούμε ότι μπορεί το ίδιο εγχείρημα να έχει θετική κατάληξη, 100% ε, θα είμαι υπέρ. Διότι θεωρώ ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την κοινή στρατηγική αντίληψη και ταυτόχρονα να προχωρήσουμε την συνεργασία μας με το ΝΑΤΟ. Αυτά είναι συμπληρωματικά, δεν είναι αντιφατικά μεταξύ τους. Ευχαριστώ. Κύριε Μπορέλα, έχετε και άλλη ερώτηση. Ερώτηση. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Εντάξει, των άλλων μέσων πολιτικής που έχουμε, έχουμε το άρθρο 42 7, όπου έχει αυτή την ρήτρα αμοιβαία βοηθεία. Ήδη έχει ενεργοποιηθεί το 15 από τη Γαλλία για τις τρομοκρατικές επιθέσεις και πολλές άλλες χώρες μέλη ανταποκρίθηκαν. Άρα θα πρέπει να αντιλήσουμε κάποια συμπεράσματα από το 42.7. Στο μέλλον να ενεργοποιείται αυτό το άρθρο και να περιβάλλεται από καλύτερο συντονισμό και ταχύτερη δράση. Επομένω, να εκμεταλλευτούμε όσο μπορούμε περισσότερο το 42 και στο μέλλον, να μπορέσουμε έτσι να αντιμετωπίσουμε τις υβριδικές απειλές για τις οποίες μιλήσατε. Εσείς συγκεκριμένα πώς τα βλέπετε. Πώς μπορούμε κάτι να κάνουμε τόσο ώστε να αξιολογήσουμε την ενεργοποίηση του 42-7. Τι ρόλο θα μπορούσε να έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν έρθει η ώρα. Μπορέλ. Έχετε το λόγο, λέει ο Πρόεδρος, κύριε Μπορέλ. Σίγουρα. Αυτό το άρθρο είναι ένα άρθρο που θα πρέπει να αποκτήσει επιχειρησιακό χαρακτήρα. Τα είπατε σε κάποια δραματική καμπή της ιστορίας της Γαλλίας. Όλοι θυμόμαστε τι έγινε. Και αυτό το άρθρο, όπως κι άλλο ένα, νομίζω το 2.12, αυτό το οποίο αφορούσε την ε, κοινή ανταπόκριση κατά αυτών των τρομοκρατικών επιθέσεων ε, για αντιμετώπιση θεομηνιών, για πάρα πολύ ε, σοβαρές περιπτώσεις, που πράγματα εκτός ελέγχου, όπως η μανία της φύσης. Οπότε θα πρέπει έτσι να εφαρμόζονται αυτά τα άρδρα και όπως ε, είπαμε έτσι διαμορφώνεται η εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Να, πώς κανείς περνά από τα λόγια στα έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μια αμυντική ένωση όπως είναι το ΝΑΤΟ. Το 42-7 είναι ό,τι πιο ε, επιχειρησιακό έχουμε και βέβαια το 212 μιλάει για στρατιωτική απειλή όλα. Τι γίνεται με την κυβερνοαπειλή δεν είναι με στενή έννοια ε, Στατιωτική φύσεω. επομένω, δεν θα ίσχυε το 2.12 αλλά το 42.7 στην περίπτωση μιας τέτοιας κυβερνοαπειλή. Ο επόμενος. ευχαριστώ για το ΕΛΚ. Ο κύριος Ντανζόν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπορέλα, στα δεξιά σας ε, με ένα θεματικό γεωγραφικό χαρτοφυλάκιο τόσο ευρύ για θέματα που αποτελούν σε μεγάλο βαθμό προνομία των κρατών τη Ένωση είναι σαν αδύνατη αποστολή σα κατά κάποιο τρόπο. Εδώ και δέκα χρόνια, δυστυχώ, και ανεξαρτήτως των προσώπων, ο απολογισμό τη Ευρωπαϊκή Δημοκρατία δεν είναι και ο, πλέον ένδοξο, και δυσκολευόμαστε να αναφέρουμε μία κρίση που εδώ και δέκα χρόνια τώρα ε, η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία θα διαδραμάτισε έναν αποφασιστικό ρόλο Κάνουμε πολλά, λίγο πολύ παντού, αλλά η εντύπωση που δίνεται είναι αυτό, του κατακαιρματισμού ε, της διασποράς των προσπαθειών. Και θα ήταν καλό, πιστεύω, κύριε Οριστέντα, είπατε εκπρόσωπε, να οριστούν κάποιες προτεραιότητες. Ορίστε εσείς για τον αυτό σα κάποιε προτεραιότητες. Σίγουρα δεν θα ικανοποιηθούμε όλοι, αλλά πείτε μας ένα θεματολόγιο, κάποιε βασικέ προτεραιότητε ε, που θα διαρθρώσετε γύρω από αυτέ τι δράσει απάντηση. Σας ευχαριστώ που περιγράφει τόσο αδύνατη την αποστολή μου. Δεν με ενθαρρύνεται και τόσο πολύ βέβαια, αλλά πρέπει να σας πω ότι όταν ήμουν μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα συζητούσαμε αυτά, συζητούσαμε αυτή τη θέση, πίστευα και εγώ ακριβώς αυτό, ότι πρόκειται για αδύνατη αποστολή. Μα ακούστε, βάστε πάρα πολλά πράγματα στο χαρτοφυλάκι ενό μόνο προσώπου. Αδύνατη ή όχι, πάντω αυτή η αποστολή είναι πάρα πολύ απαραίτητη και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να το εφαρμόσουμε. Ξέρετε τι λέμε στα ισπανικά, το κάναμε γιατί δεν ξέραμε ότι ήταν αδύνατο, ότι ήταν ανέφικτο. Σας άκουσα σε ένα βίντεο στο YouTube και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε εκεί. Είπατε κάποια πράγματα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και συμμερίζομαι απόλυτα τις απόψεις σας. Πρέπει να έχουμε μια συμπληρωματική ε, στρατηγική ε, δυνατότητα και φυσικά δεν μπορούμε να είμαστε παντού, αυτό είναι σαφές, γιατί πολλές φορές δεν έχουμε την ίδια δυνατότητα ικανότητα δράσης. Τώρα, τις προτεραιότητες. Είναι δύσκολο το ερώτημα. Διότι ό,τι και αν πω, κάποιος θα δυσαρεστηθεί, θα μείνει παραπονεμένος. Αλλά αφού το ζητάτε, τα Βαλκάνια, νομίζω ότι πραγματικά και τα ανατολικά σύνορα είναι οι προτεραιότητες ε, της εξωτερικής μας πολιτικής. Δεν θα είμαστε γεωπολιτικοί αν δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα της άμεσης γειτονία. Και αν μου επιτρέπετε, και η Λιβύη είναι κάτι προφανές. Ε, ξέρω ότι δεν υπάρχει ακόμη ενότητα μεταξύ των Ευρωπαίων, αλλά ίσως να μην αντιλαμβανόμαστε ακόμη τι τεράστια απειλή είναι μια αποσταθεροποιημένη Βόρεια Αφρική. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα εδώ και αν δεν το καταφέρουμε δύσκολα θα μπορέσουμε να διαδραματίσουμε τον ιονδήποτε ρόλο ε, στην παγκόσμια ισορροπία μεγάλο πράγματι και ευρύ το πεδίο, αλλά βασίζουν και στη δική σας βοήθεια για να μπορέσει να αποφέρει κάποιους καρπούς η προσπάθειά μου. Ευχαριστώ. Ο Αρνό για συμπληρωματική, Αρνό Ντανζάν παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπορέλ, σας ευχαριστώ για την καλή απάντηση, αν μου τρέπετε. Λοιπόν, όπως και εσεί έτσι και εγώ πιστεύω ότι ε, αν δεν μπορέσουμε στην άμεση γειτονία να προασπίσουμε τις αξίες μας, δεν θα μπορούμε να αναλάβουμε παγκόσμια αποστολή. Ε, σας πηγαίνω λίγο πιο μακριά στο Σαχέλ. Μιλήσατε για τη Βόρεια Αφρική, εγώ σας πάω στο Σαχέλ και είπατε εσείς ε, ότι έχουμε όλους αυτούς τους άνδρες γυναίκες που υπηρετούν σε στρατιωτικές και μη στρατιωτικές αποστολές. Εδώ μιλάμε για μεγάλη πρόκληση στο δόμο της ασφάλειας και της ανάπτυξης. Εδώ και 10 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση φτιάχνει στρατηγικά σχέδια, ανακοινοθέντα ε, που εντοπίζουν τα προβλήματα και ζητούνται λύσει. Δυστυχώ όμω η δράση μα δεν φαίνεται αποφασιστική. Ε, ποια είναι η δική σα άποψη, τι προσοχή θα δώσετε στην περιοχή αυτή, τι δράσει μπορούν να αναλυφθούν. Πράγματι, εγώ πήγαν σε Νίγηρα, σε Νεγάλη και πράγματι δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι το Σαχέλ για την Ευρώπη είναι το νότιο σύνορο ουσιαστικά σε Ευρώπη Οι Άραβες ε, χρησιμοποιεί τη λέξη φύτα που περιγράφει αυτά που γίνονται. Ουσιαστικά μία μόνιμη αντιπαράθεση δομική ε, μεταξύ οικονομικών παραγόντων, ε, καλλιεργητών της γης, γεωργών κτλ. Πρέπει να δεσμευτούμε, να ασχοληθούμε πολύ περισσότερο, γιατί δεν είναι μόνο λίκνο της τρομοκρατίας ενίοτε, αλλά από εκεί μπορούν να αναδεθούν πάρα πολλές γεωστρατηγικές απειλές. Μιλάμε για 200 εκατομμύρια κατοίκους. Θα πρέπει να έχουμε ένα πράσινο σύνορο, αν μπορώ να το πω έτσι. Αυτό το ζήτησαν οικολόγοι, για να μην επεκταθεί έρημος ε, της Σαχάρας. Θέλουμε ε, επιμόρφωση, δημιουργία υποδομών, βοήθεια της δημόσιας διοίκησης. Ε, πράγματι λοιπόν είναι και αυτή μια προτεραιότητα. Ευχαριστούμε. Υποψήφια είπατε εκπρόσωπε. Περνάμε στον επόμενο μιλητή μας, Σβέν Μίξερ από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Κύριε υποψήφια, θα ήθελα να επανέλθω σε θέματα άμυνας και ασφάλειας ε, και να περάσω στις ε, πραγματικές ικανότητες όταν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας ε, και την διαρθρωμένη συνεργασία. Θεωρώ ότι αφενός ο ρόλος αυτών των προτεραιοτήτων είναι να ισχύσουμε τις κοινέ μας προσπάθειες και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά μας στον τομέα της στρατιωτικής βιομηχανίας, αλλά από την άλλη και ευρύτερα ο στόχος είναι να έχουμε στην διάθεσή μας τις απαραίτητες δυνατότητες για να ανταποκριθούμε στις διεθνείς μας υποχρεώσεις και τις φιλοδοξίες που αναφέρει η παγκόσμια ατζέντα μας. Οπότε το ερώτημά μου είναι το εξής. Πού βλέπετε να υπάρχουν μεγαλύτερες ελλείψεις ε, και πώς σκοπεύετε να εργαστείτε και στο επίπεδο της Ένωσης και με τα κράτη στο διακυβερνητικό επίπεδο για να αντιμετωπιστούν αυτές οι ελλείψεις. Κύριε Μπορέλ, για δύο λεπτά. Θα προσπαθήσω να απαντήσω αυτή τη δύσκολη ερώτηση σε δύο λεπτά. Συγκεκριμένα, πρώτα απ' όλα, συμφωνήσαμε σε ένα σχέδιο ανάπτυξης ε, δυνατοτήτων ε, που έχει 11 προτεραιότητες για την άμυνα. Αυτές περιλαμβάνουν, το γνωρίζουμε, τις ε, κυβερνοεπιχειρήσεις, ανεφοδιασμό στον αέρα και, άμυν, και βαλιστική άμυνα. Ε, θυμάστε ότι όταν γίνονταν πλήγματα στην Λιβύη δεν μπορούσαμε να ανεφοδιάσουμε τα αεροσκάφη μας και χρειαστήκαμε τη βοήθεια των Αμερικανών. Κατόπιν, οι ικανότητε αυτές είναι κάτι που χρειαζόμαστε για τις επιχειρήσεις ΚΕΠΑ. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, και την συμβατότητα και συμπληρωματικότητα με το ΝΑΤΟ. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η έχουν έναν τύπο άρματος μάχης. Εμείς έχουμε 17 ε, διαφορετικούς τύπους. Η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των ε, κρατών μελών στον τομέα αυτών μας κοστίζει ε, γύρω στα 30 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πρέπει να αναπτύξουμε την ΚΕΠΑ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Είναι πολύ φτηνότερο να ξοδεύουμε σε συνεργασία από το να έχουμε πολλές διαφορετικές ικανότητες ασύμβατες μεταξύ τους και πολύ ακριβές. Πρέπει επίσης οι πόροι να ανταποκρίνονται στις φιλοδοξίες. Και το πει εκεί υπάρχει, εσείς πρέπει να αποφασίσετε. Και πρέπει να δούμε και την πολιτική διοίκηση που είναι εξίσου σημαντικό για εμένα όσο οι στρατιωτικές αποστολές και για το λόγο αυτό χρειαζόμαστε άλλες δυνατότητες ε, αστυνομικούς, δικαστές, εισαγγελείς ε, και τα λοιπά. Σας ευχαριστώ. Α, άλλη ερώτηση. Ε, ευχαριστώ. Συμφωνώ ότι η συνεργασία είναι η λέξη κλειδί αλλά έχουμε δει και στο παρελθόν περιπτώσεις όπου καταφέραμε να συνεργαστούμε για να υποδομηθεί κάποια δυνατότητα η οποία τελικά παρέμεινε χρησιμοποιητή, παραδείγματος χάρη οι ομάδες μάχης. Θεωρώ λοιπόν ότι οι ομάδες αυτές έχουν κάποια αξία ε, στην υπόθεση αυτή του μετασχηματισμού, αλλά δεδομένων των περιορισμών οικονομικών και πολιτικών που βλέπουμε. Πώς θεωρείτε ότι θα αντιμετωπίσουμε αυτούς τους περιορισμούς για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που θα έχουμε από κοινού. Ευχαριστώ. Κύριε Μπορέλ. Ναι. Οι διάσημες αυτές ομάδες μάχης που δεν χρησιμοποίησαν ποτέ. Παρ' όλα αυτά, παραμένουν το βασικό εργαλείο ταχείας αντίδρασης και είναι οι μόνες ε, δυνάμεις που έχει έτοιμες η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να τις αναπτύξει. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να αυξήσουμε την κοινή μας χρηματοδότηση που συζητείται αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου Ειρήνης ε, που πρότεινε η κυρία Μογκερίνη για να υπάρξει ακριβώς ένα κίνητρο για μελλοντικές αναπτύξεις έτσι ώστε όταν είχε έρθει η στιγμή, θυμάστε η περίπτωση με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και το Μαλί, δεν θέλω να ασκήσω κριτική τώρα, αλλά για διάφορους λόγους δεν υπήρξε κινητοποίηση. Λοιπόν, αν υπάρχουν αυτές οι ε, μονάδες μάχης, πρέπει να υπάρχει κοινή χρηματοδότηση, γιατί είναι τα εργαλεία της ευρωπαϊκής στρατιωτικής δυνατότητας. Ευχαριστούμε περνάμε στον επόμενο μιλητή, τον Πρασίνο, η κυρία Γενμπού. Παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Κύριε Μπορέλ, λέτε ότι πρέπει να είμαστε συνεκτικοί και συνεπείς σε διεθνές επίπεδο και συμφωνώ. Αλλά καλύτερα να ξεκινήσουμε με, από τα του οίκου μας. Λέτε ότι είστε πεπισμένος φεμινιστής εδώ και χρόνια. Πώς λοιπόν συγκεκριμένα και επιμένω θα φροντίσετε κεφαλή της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας ε, να ε, έχει πιο έτσι, γυναικεία χαρακτηριστικά. Το 75% της ΕΕΔ ε, στα, μέσα στελέχη είναι άντρες ε, και σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο προσωπούνται στα ανώτερα στελέχη, πάνω από το 80%. Πώς θα προωθήσετε την ισότητα των φίλων στην παρουσία γυναικών, δηλαδή τουλάχιστον 50% μέχρι το 2024 να είναι γυναίκες επικεφαλής στις διάφορες αντιπροσωπείες ψηφίσει στο Κοινοβούλιο και τι θα κάνετε με τις λιγότερο ευνοημένες ομάδες πληθυσμού. Δυστυχώς η διπλωματία πολλές φορές είναι συνώνυμο της κοινωνικής πολιτικής ελίτ. Τι θα κάνετε για να αλλάξει αυτό, να υπάρχει περισσότερη ισότητα στο χαρτοφυλάκιό σας. Ευχαριστώ ένα λεπτό, μάλλον δύο λεπτά, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος, κύριε Μπορέλ. gender equality is... Η ισότητα των φύλων θεμέλιο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η πρόεδρος Φαντερ Λάιν το είπε ξεκάθαρα. Η ισότητα των φίλων στην εξωτερική πολιτική δεν σημαίνει μόνο η εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στις υψηλές θέσεις. Ήδη έχουμε γύρω στο τρίτο γυναίκε. Για να είμαι ειλικρινή, νομίζω ότι θα είναι αδύνατο να φτάσουμε το 50% στο χρονοδιάγραμμα που προτείνεται. Μπορώ να πω ναι, αλλά προτιμώ να είμαι ειλικρινή. Θα λέγω ότι ένα καλός στόχος είναι γύρω στο 40% να θυμάστε ότι το 1 τρίτο των θέσεων της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης ε, μας το δίνουν οι εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες που έχουν και αυτές ανάλογες απαιτήσει. Οπότε υπάρχει εδώ πέρα μια σύγκρουση για α, σπάνιους πόρους που είναι αυτή τη στιγμή οι γυναίκες με προσόντα στο διπλωματικό σώμα. Έχω αυτή τη συζήτηση και στο εσωτερικό. δεν ξέρω αν θα είναι βραχυπρόθεσμα δυνατό το 50% αλλά κάτι πιο σημαντικό ή εξίσου σημαντικό είναι να μπουν τα θέματα του φίλου στις ε, διπλωματικές και στρατιωτικές δραστηριότητες στο εξωτερικό. Δεν έβλεπα έναν συνταγματάρχη του στρατού του Μαλή που εξηγούσε τον ρόλο των γυναικών σε τέτοιες συγκρούσεις. Δηλαδή έλεγε ότι το ότι ήταν γυναίκες στο στρατό ε, ήταν ο μόνος ε, τρόπος ε, να εμπιστευτούν οι γυναίκες οι άλλες τον στρατό που τις βιάζανε λοιπά. Πρέπει λοιπόν να ενσωματωθεί αυτό στις πολιτικές και στρατιωτικές δραστηριότητες. Θα έχετε και άλλη ερώτηση κυρία Γεμπού. Συμφωνείτε με το ότι είναι ντροπή η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που γίνεται με το άσυλο δεν θα πρέπει να καταγγελθεί η κατασκοπή από την Υπηρεσία Ασφαλείας των Πολιτειών. Αυτό είναι κινησμός και υποκρισία. Δεν θα πρέπει να έχουμε κοινή θέση. Δεν θα πρέπει να ξεμπλοκαριστούμε. Εσείς δεσμεύεστε να πείσετε τους Αγίους Καρνό και Κυβερνήσεων να αναθεωρήσουν το τι έγινε με τον Σνόντεν όταν ζήτησε άσυλο. One Για ένα λεπτό, κύριε Μπορέλ. Κυρία ε, βουλευτή, πώς να σας απαντήσω. Δεν έχω την αναγκαία ενημέρωση, ούτως ώστε να γνωρίζω τι είναι αυτό, ποια είναι η απάντηση στο ερώτημά σας. Δεν γνωρίζω είναι η ειλικρινή απάντησή μου. Thank you. Ευχαριστούμε λίγο Πρόεδρο. Ομάδα ID Patrick Berg. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μπορέλ, στις γραπτές απαντήσεις σας λέτε ότι σκοπεύετε να εκμεταλλευτείτε πλήρως τις δυνατότητες της συνθήκης της Λισαβόνας για να περάσουμε σε ψηφοφορία με ε, διευρυμένη πλειοψηφία, με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Μπορείτε να μας πείτε ποιοι τομεί θα ήταν κατάλληλοι για ειδική πλειοψηφία και μπορείτε να μα πείτε αν αυτό αποτελεί διάβρωση τη εθνική κυριαρχία. Λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λαμβάνει αποφάσει γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα. Και πρέπει οι περιορισμοί αυτοί να ξεπεραστούν που εμποδίζουν την εξωτερική μας πολιτική. Εννοείται δηλαδή ότι οι διαφορές απόψεων είναι κατά της κοινή εξωτερικής πολιτικής και θέλω να αναφερθώ και στην, στα θέματα της ε, μεταναστευτικής. Μπορεί βεβαίως με τα ανθρώπινα δικαιώματα να είμαστε προς το συμφέρον ε, των μεταναστών, αλλά είναι προς το συμφέρον των πολιτών της Ευρώπης. Πρόκειται για μια απειλή ασφαλείας ή όχι. Σας ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Κύριε Μπορέλ, δύο λεπτά. Πραγματικά ε, είναι δύο αυτά που με ρωτήσατε. Να σας πω σε δύο λεπτά αν γίνεται. Το προείπα για εμένα είναι κάπως αντιφατικό το να ε, έχουμε απέτηση ομοφωνίας στα οικονομικά, στις δημοσιονομικές προοπτικές, όπου συζητάμε το 1% του ΑΕΠ και απαιτούμε ομοφωνία και μετά θέλουμε να λαμβάνουμε αποφάσεις πολύ πιο σημαντικές που αφορούν, όπως είπα, ανθρώπινα δικαιώματα, πόλεμο και ειρήνη, με ειδική πλειοψηφία. Θα ήταν πολύ πιο απλή η δουλειά μου, εάν ε, είχαμε ειδική πλειοψηφία. Αλλά δεν μπορούμε να επιβάλλουμε μία απόφαση σε ένα κράτος μέλος παρά τη θέλησή του, όταν αφορά τόσο σημαντικά πράγματα. Ας τα πάμε βήμα-βήμα. Ας ξεκινήσουμε με την ειδική πλειοψηφία στις ε, κυρώσεις, όπως στην περίπτωση της ε, Ρωσίας, να μην χρειάζεται ομοφωνία, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις ειρηνευτικές αποστολές. Και μετά μπορούμε να έχουμε αυτή την κοινή κουλτούρα για να συμφωνήσουμε σε τέτοια ζητήματα που αφορούν την κυριαρχία. Ε, δεν έχουμε την... Αν δεν έχουμε την ίδια αντίληψη δεν μπορούμε να έχουμε κοινή εξωτερική πολιτική. Πόσο καιρός χρειάστηκε για να πάμε από το κοινό νόμισμα στο ενιαίο νόμισμα. Για να πάμε από την ε, μοιρασμένη ε, κυριαρχία στο να έχουμε τελικά ένα νόμισμα το οποίο οπωσδήποτε ήταν εγκατάλειψη ή μάλλον διαμοιρασμός της ε, εθνικής κυριαρχίας. Πρέπει να πάμε Βήμα-βήμα λοιπόν, αλλά ο τελικός στόχος είναι οι αποφάσεις να λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία όταν θα έρθει η ώρα. Ευχαριστώ. Έχετε κι άλλη ερώτηση κύριε συναδελφοί. Το δεύτερο κομμάτι της ερώτησής μου αφορά την ε, δίωξη χριστιανών ανά τον κόσμο. Είχαμε μία έκθεση της είπα της εκπροσώπου για την Μπουρκίνα Φάσο όπου είχαμε συστηματικές ε, διώξεις των χριστιανών και νέες εκκλησίες και τα λοιπά. Αυτό είναι πολύ διαδεδομένο στο Σαχέλ, Μέση Ανατολή και Αφρική. Και ένα από τα πολλά παραδείγματα των τελευταίων ετών. Εδώ υπάρχει μια έντονη στήριξη για πρόταση διαφόρων μειονοτήτων, αλλά σχεδόν καμία για τους χριστιανούς. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι πολύ δημοφιλές ε, κάτι τέτοιο, αλλά δεν ξέρω, ελπίζω, νομίζω ότι συμφωνούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε κάποιες ευρωπαϊκές αξίες και θα έπρεπε να υπερασπιστούμε τους χριστιανούς. Ανησυχεί η Κομισιόν για την αυξανόμενη βία κατά των χριστιανών και τι σκοπεύει να κάνει γι' αυτό. Σας ευχαριστώ κύριε Μπορέλ. Δεν ξέρω λοιπόν αν είναι διαδεδομένο ή όχι, αλλά συμφωνώ μαζί σας ε, γιατί βεβαίως η ανεξαρτησία είναι ε, θεμέλιο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Δηλαδή, για, κάναμε πολέμους ε, θρησκευτικούς, η ανεξαρτησια ειναι ε θεμελιο του ευρωπαικου πολιτισμου πόλεμη, ε, κάτι το οποίο προκαλούσε λουτρά αίματο ε, στην Ευρώπη για πολλούς αιώνε και τώρα σεβόμαστε όχι μόνο του χριστιανούς αλλά τους πάντες και ξέρω πολύ καλά το τι συμβαίνει ε, στην Μπουρκίνα Φάσο και στο Ιράκ ε, όπου καταστρέφονται και διώκονται συνεχώς οι κοινότητες χριστιανών. Οπωσδήποτε λοιπόν πρέπει το θέμα αυτό να το δούμε ε, σε όλες τις πτυχές της εξωτερικής πολιτικής μας. Και η Μπουρκίνα Φάσο είναι στο πλαίσιο αυτής της ε, θέτα που λέμε. Ε, η γενικευμένη βία πάντων κατά πάντων στο ε, ήταν πολύ πιο έντονη η κατάσταση. Σας ευχαριστώ για το ECR Hammond Hertz. Για ένα λεπτό. Καλησπέρα κύριε Μπορέλ και καλώς ορίσατε στο Κοινοβούλιο που το ξέρετε καλά. Εδώ, εδώ είναι. Λέει ο κύριος Εγώ θα σταθώ και πάλι στο θέμα των κυρώσεων. Εσείς δεν πιστεύετε στις κυρώσεις. Αν είχαμε τη θέση που είχαμε υιοθετήσει για Βενεζουέλα και Κούβα, γιατί και αυτό θα πρέπει να το δούμε, τότε αν είχαμε τη θέση αυτή για, για Ισραήλ και Κούβα, εδώ είχαμε και για Νοτιοαφρικανική Δημοκρατία και μιλάμε για 25.000 άτομα, 25 άτομα συγγνώμη, που είναι τώρα αποκλεισμένοι στη Βενιζόλη λόγω και έχουμε επίση 5.000 ε, πρόσφυγες Βενζολάνους 5 εκατομμύρια συγγνώμη οι οποίοι φεύγουν από το καθεστώς για να γλιτώσουν και άρα είναι 25, ξαναλέω, μιλήσει Ευρωπαίοι, οι οποίοι τώρα είναι αποκλεισμένοι στην ε, Βενεζουέλα και κανεί στην Κούβα. Έχετε δύο λεπτά, κύριε Μπορέλ. Ευχαριστώ, κύριε Δεν είπα ότι είμαι κατά των κυρώσεων. Είπα ότι είμαι κατά των συλλογικών ενεργειών που αρνητικά επηρεάζουν τον λαό της Βενεζουέλας. Όταν κανείς γνωρίζει την εκεί κατάσταση, ό,τι εμποδίζει το να μην έχει ο κόσμος φάει να φάει είναι κάτι που με βρίσκει αντίθετο. Και το είπα στους Αμερικανούς φίλους, ας μην υποστηρίξουμε συλλογικές κυρώσεις κατά του λαού. Ναι, ατομικές κυρώσεις κατά των αξιωματούχων. Εμείς το κάνουμε αυτό στην Ισπανία κατά επτά αξιωματούχων που έκαναν ε, εγκλήματα στα πλαίσια του ναυτικού της χώρας στη Βενεζουέλα. Και προς τα εκεί, προς αυτή την κατεύθυνση προσπαθούμε τόσο ώστε να βρεθεί η καλύτερη λύση. Η καλύτερη λύση με διαπραγματεύσεις μεταξύ ε, των αντιπαρατεθειμένων των διαφόρων μερών στη χώρα και δεν είναι το θέμα μόνο θα γίνει με την Κούβα, είναι και άλλες ε, χώρες, είναι τα πράγματα πιο περίπλοκα από ό,τι φαίνεται. Είμαι κατά όχι των κυρώσεων, των συλλογικών τιμωριών και κυρώσεων που χτυπάνε τον λαό που ήδη και σε δραματική κατάσταση και για την Κούβα. Κοιτάξτε, εσείς εγκρίνετε και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια μέτρα απομόνωση της Κούβας. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Κανένα αποτέλεσμα και μετά από λίγα χρόνια υπήρξε συμφωνία και ακόμα και ο Πάπας συνέχισε τις σχέσεις με την ε, χώρα. Η Γαλλική Δημοκρατία και όχι ο βασιλεύς της Ισπανίας. Ε, αυτό έγινε. Σας ευχαριστούμε, λέει. Ο πρόεδρος επερώτηση. Έχετε κύριε Τέρτσου, για ένα λεπτό. να παρουσιάζετε ε, την κούφα φυσιολογική χώρα που πάνε όλοι, ενώ που πραγματικότητα είναι ένα κελί, μια φυλακή ε, που υποστηρίζει το καθεστώ στη Βενεζουέλα και έχουμε 5 εκατομμύρια από τη Βενεζουέλα, 1 εκατομμύριο στην Κολομβία που έχουν φύγει ε, τι να μας λέτε ότι είναι φυσιολογική υπέροχη χώρα, δεν νομίζω. Ε, δεν είναι θέμα μέτρων. Ε, είναι το θέμα πώς θα χτυπήσουμε την τελευταία κομμουνιστική δικτατορία που αποσταθεροποιεί το, το ημισφαίριο αυτό. Δεν είπα ότι είναι υπέροχη τέλεια χώρα. Νομίζω ότι μιλούμε την ίδια γλώσσα εσείς και εγώ. Δεν είπα ότι είναι υπέροχη η Κουβά, είπα ότι από εκεί περνούν ότι εκεί πάνε όλοι. Είναι αλήθεια ή όχι. Ισχύει ή όχι. Ο Ομπάμα δεν πήγε, ο Πάπα δεν πήγε, δεν πήγε ο πρόεδρος Γαλλική Δημοκρατία. Μόνο εμεί δεν πήγαμε. Η μόνη κομμουνιστική δικτατορία που έμεινε στον κόσμο, είπατε, είστε σίγουροι γι' αυτό. Ο Ραλου Κάστρο μια μέρα ξέρετε τι είπε. Μου είπε, εμένα να με μεταχειρίζετε σαν να ήμουν Σαουδάραβας, Κίνα, Κινέζος κλπ. Ναι, έχουμε αυτή την ε, φιλοδοξία να έχουμε σχέσεις με τους φίλους λαούς. Όχι, δεν κανένας κατευνασμός. Έχουμε πολιτική επαφών που αφήνει περιθώριο για σχέσεις λαών και κυβερνήσεων. Όχι στην πολιτική απομόνωση που δεν οδηγεί σε τίποτα. Ευχαριστώ. Από το ΕΛΚ, η κυρία Ιζαμπέλ Λίμα. Να έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπορέλ, εδώ είμαι. Η ε, ελευθερία έκφραση και λόγου, ο πλουραλισμό των μέσων ενημέρωση είναι στο επίκεντρο των αθεκτικών δημοκρατικών κοινών και πρέπει να προστατεύσουμε αυτά τα στοιχεία. Τι προστατευτικά μέτρα θα εφαρμόσετε για να αντιμετωπίσετε τις εκστρατείες παραπληροφόρησης ε, και την εχθρική καμπάνια απ' έξω προς ε, την Ένωση και τα κράτη-μέλη της. Αναφέρθηκε ήδη τρομοκρατία που πλήττει τις ατομικές ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών σε όλο τον κόσμο. Η δική σας θέση ποια είναι σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας που συχνά είναι απαραίτητο να εφαρμόσουν οι χώρες που ενδεχομένως όμως περιορίζουν τελικά και τις ελευθερίες. Αυτή τη στιγμή πολλοί ε, πολιτικοί και άλλοι ακτιβιστές αγωνίζονται για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Και συχνά είναι, προ... Ε, αντικείμενο εκφοβισμού, ίσως και χάνουν τη ζωή τους, δολοφονούνται το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, πώς θα τον συμπεριλάβετε πέραν των οικονομικών σχέσεων και στις άλλες διεθνείς επαφές και σχέσεις που έχετε. Ευχαριστώ. Απάντηση. Νομίζω ότι με κάποιο τρόπο έχω ήδη απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τις δυνατότητες που έχει. Ουσιαστικά πρόκειται για τις διπλωματικές σχέσεις και την άσκηση πολιτικής πίεσης Ιδίω στις χώρες εκείνες που δεν συμμορφούνται προς τα πρότυπα και τους κανόνες που απαιτούμε εμείς. Αναφερθήκατε στο πολύ σοβαρό πρόβλημα τη παραπληροφόρησης. Αυτό δεν αφορά μόνο τη Ρωσία, αλλά σε μεγάλο βαθμό την αφορά. Και είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχήσει. Όχι, ναι. Ορίστε. Εγώ δεν αναφέρθηκα στη Ρωσία, δεν κατονόμασα. Εγώ το κάνω, Λίκρος Μπορέλ. Εγώ ναι, το λέω. Λέω. Το ξέρουν όλοι στον κόσμο ότι υπάρχουν στρατές παραπληροφόρησης από σερβερ ε, που βρίσκονται σε ε, ρωσικό έδαφος. Δεν ξέρω τι δεν λέω ότι είναι η ε, ρωσική κυβέρνηση. Sputnik και Ράσια του Ντέιν είναι ιδιωτικέ επιχειρήσει, λέει ο κ. Λαυρόφ, αλλά υπάρχουν εκστρατείες παραπληροφόρησης ε, που πλήττουν την δημοκρατική ευρωστία, την δημοκρατική υγεία των χωρών μας και η παραπληροφόρηση πρέπει να είμαστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε ως ένα από τα βασικά στοιχεία και της τεχνητής νοημοσύνης. Θα αποδυναμώνει τις διαδικασίες που βασίζονται στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα μέχρι τώρα. Έχουμε τα στραντς. τρία. Ένα αφορά την Ανατολική Ευρώπη, Έχουμε το σώμα γρήγορης αντίδρασης κατά της παραπληροφόρησης, περιορισμένη δυνατότητα παρέμβασης. Άρα θα πρέπει να έχουμε πολύ περισσότερες δυνατότητες γιατί το πρόβλημα θα επιδεινούται όσο περνάει ο χρόνος. Γιατί τα τεχνολογικά εργαλεία και μέσα τα οποία αναπτύσσονται δυστυχώς διακόπτεται ο κύριος Μπορέλ. Ευχαριστώ. Επερώτηση. Κύριε Μπορέλ, Με ικανοποίησε απάντησή σα, αλλά θα ήθελα μια διευκρίνηση συγκεκριμένα σε σχέση με αυτό που υπόθηκε πριν. Η ελευθερία λόγου πηγαίνει μαζί με την ελευθερία πεποίθηση, πιστεύω, τη θρησκευτική ελευθερία, τη δικαίωμα να μην έχει κανείς ε, πίστη σε κάποιο δόγμα. Και υπάρχουν πολλές συγκρούσεις ε, και πόλεμοι λόγω όλων αυτών. Εσείς συγκεκριμένα πώς δεσμεύεστε σε σχέση ιδίως με το Global Exchange on Religions and Society, μια πλατφόρμα από ε, την αγίδα της Ένωσης που δρομολόγησε είπατε εκπρόσωπος, εσείς τι θα κάνετε σε σχέση με αυτή την πλατφόρμα για να προστατεύσετε τις θρησκευτικές μειονότητες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς θα βελτιωθεί ε, και το περιθώριο του ειδικού απεσταλμένου για αυτά τα θέματα. Και τέλος, παντού στον κόσμο η ανισότητα ανδρών και γυναικών ε, είναι διαδεδομένη. Η νομοθεσία δεν προστατεύει συχνά. Εμείς είμαστε προσιλωμένοι στην αρχή της ισότητας. Πώς θα την προωθήσουμε σε όλες τις υπήρους την ισότητα. Ευχαριστώ. Κύριε Μπορέλ, έχετε ένα λεπτό. Ε, τελικά θα με πείσετε ότι είναι αδύνατη η αποστολή που έχω αναλάβει. Πώς θα λύσω εγώ το πρόβλημα της ισότητας των φίλων σε όλες τις υπήρους. Ε, τι να σας πω. Εγώ γνωρίζω την πρωτοβουλία αυτή της κυρίας Μογκερή, αυτή την πλατφόρμα που αναφέρατε και την υποστηρίζω και θα προσπαθήσω να την προωθήσω για τον πολύ απλό λόγο ότι είμαι ένας άνθρωπος κοσμικός, πιστεύω δηλαδή στην κοσμίκευση και πιστεύω και στην ε, ελευθερία θρησκεία, θρησκευτική ελευθερία που πρέπει να προστατευτεί. Γιατί υπάρχουν πολλέ χώρε που δεν είναι σεβαστή θρησκευτική ελευθερία. Το είδαμε και σε κάποιε άλλε ερωτήσει συναδέλφων σα. Άρα η πρωτοβουλία τη κυρία Μόγκερ είναι πολύ πρόσφατη, από το Σεπτέμβριο, κανένα μήνα έχει περάσει, από τότε που δρομολογήθηκε, νομίζω ότι είναι κάτι που πραγματικά πρέπει να αναπτυχθεί και εγώ προσωπικά εκπεπιθήσεως, εκφύσεως, ε, θα την υποστηρίξω. Είναι κάτι φυσικό για μένα. Ευχαριστώ. Thank you, ευχαριστώ. Περνάμε στον επόμενο μιλητή. Από την ομάδα New Europe, Urmas Σας ευχαριστώ κύριε Μπορέλ. Ε, λίγο πολύ συμφωνούμε ότι οι γείτονε μας έχουν ε, σημασία και η ανατολική γειτονία είναι προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης καθώς πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει την ασφάλεια και την σταθερότητα στα σύνορα της όμως η Ρωσία συνεχίζει να εισβάλλει στην Ουκρανία, Ντον Μπάς, Μολδαβία, Απχαζία, Νότια Οσετία και απειλεί και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς σκοπεύετε λοιπόν να διατηρήσετε ως προτεραιότητα την ανατολική γειτονία, λαμβάνοντας υπόψη ε, και τα απαραίτητα οικονομικά μέσα στον ε, ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και τι ακριβώς σκοπεύετε να κάνετε για να συμμεθεί κάποια πρόοδο στην επίλυση αυτών των συγκρούσεων στις χώρες αυτές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μπορέλ, για δύο λεπτά. Κοιτάξτε, ο καλύτερος τρόπος ε, για να αντιμετωπίσουμε ας πούμε, τον ρωσικό επεκτατισμό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, η ρωσική απειλή, άμα θέλετε, είναι να βοηθήσουμε την Ουκρανία, να ενισχύσουμε την Ουκρανία. Την αντοχή της, την δυνατότητά της να κάνει μεταρρυθμίσεις και να γίνει ε, μια δημοκρατική και ευμερούσα χώρα. Οι κυρώσεις ε, προς τη Ρωσία θα βοηθήσουν, αλλά νομίζω πως οι κυρώσεις δεν πρέπει να θεωρούνται ως πολιτική από μόνες τους. Είναι ένα εργαλείο και η Ανατολική Σύνδεση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως κάτι το οποίο στρέφεται κατά κάποιο. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε έναν δακτύλιο δημοκρατικών χωρών μεταξύ ημών και Ρωσίας ε, για να υπάρξει μια ισορροπημένη εφαρμογή των πέντε κατευθυντηρίων αρχών που προβλέπουν επί τη κυρία ευελιξία ε, για ρύθμιση και μικρορυθμίσεις όπου αυτό απαιτείται. Συνοψίζοντας λοιπόν, η Ουκρανία παραμένει βασικό κομμάτι της στρατηγικής πρόκλησης ας πούμε που αποτελεί η Ρωσία και είναι ε, μια βασική προτεραιότητα για να έχουμε μια αξιόπιστη εξωτερική πολιτική. Πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε αυτούς τους ε, στόχους και ξέρω βεβαίως πως ε, δεν έχει αυτό την ίδια σημασία σε όλα τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να είμαι ειλικρινής. Πρέπει να επιμείνουμε σε αυτήν την θέση και αν δεν μπορούμε να είμαστε ενωμένοι και ε, υπενθυμίζω ότι απαιτείται ομοφωνία τότε θα έχουμε πρόβλημα. Εμείς θα έχουμε πρόβλημα. Οπότε η πρώτη μου προσπάθεια θα είναι να συνεχίσουμε με την ενότητα αυτή, να αυξήσουμε την στήριξή μας στις χώρες της ε, γειτονίας. Επαναλαμβάνω και πάλι δεν στρέφεται κατά κάποιον. Σας ευχαριστώ. Θα μας πάει. Θα έχετε και άλλη ερώτηση. Ναι. Η Ρωσία έχει παραβιάσει επανειλημμένο το διεθνές δίκαιο και συνεχίζει να έχει συγκρούσεις με τις γειτονικές χώρες. Γεωργία, Ουκρανία, και ω εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες δημοκρατικέ χώρε επέβαλαν κυρώσει στη Ρωσία. Συμφωνώ ότι η συνένεση είναι σημαντική, αλλά έχετε κάποια πιο συγκεκριμένα σχέδια για το πώ θα διατηρηθεί η συνένεση μεταξύ των κρατών μελών. Και επίση τι άλλες μεθόδους ε, θεωρείτε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να επηρεάσει τα κράτη-μέλη που παραβιάζουν το διεθνές δικαίωμα να σταματήσουν να το κάνουν και ποια είναι η θέση σας για μια ευρωπαϊκή λίστα Μαγνίτσκι, παραδείγματο χάρη. Σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό κύριε Μπορέλ. Νομίζω ότι ήταν ο Θεόδωρος Ρούσβελτ που είπε ότι ε, καλό είναι να μιλάς ε, ήρεμα με ένα μεγάλο ματσούκι όμως. Οπότε, αν δεν έχεις έτσι μεγάλο ματσούκι, καλό είναι να μην φωνάζεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει. Δεν ε, έχει στρατό. Και όπως σας είπα, Πρέπει να είμαστε σκληροί με τη Ρωσία, αλλά ταυτόχρονα να αντιληφθούμε ότι είναι κάποιος με τον οποίο πρέπει να είμαστε σε επαφή. Δεν λύνονται τα πάντα με κυρώσεις επικυρώσεων. Διατηρηθούν οι κυρώσεις, αλλά ταυτόχρονα έχουμε διπλωματικά εργαλεία και την πέμπτη αρχή που μας δίνει τη δυνατότητα μιας επιλεκτικής επαφής για να ξεκινήσω ο απαραίτητος διάλογος. Σας ευχαριστώ. Από τους μη εγγεγραμμένους Nathan Gill. Στην αρχική σας δήλωση είπατε ότι η ισχυρή πολιτική απαιτεί ισχυρή δημοκρατική στήριξη. Επίσης είπατε στις 22 Μαΐου όταν σας ρώτησαν τι θα παραδίνατε πιο δύσκολα, νόμισμα ή εξωτερική πολιτική και απαντήσατε. Γεγονός είναι, το νόμισμα και τα σύνορα είναι δύο βασικά στοιχεία ενός κράτους. Δεν το αναγνωρίζουν μόνο οι Βρετανοί αυτό. Εκατομμύρια άνθρωποι σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θέλουν να παραδώσουν το νόμισμα και τα σύνορά τους και τους εθνικούς στρατούς τους που υπερασπίζονται αυτά τα σύνορα. Θεωρείτε ότι οι Πολωνοί θα παραδώσουν το σλότι ή οι Δανείοι την κορώνα. Θέτω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα σύνορα και το νόμισμά της είναι τώρα το εθνοκράτος και πώς θα έχετε δημοκρατική στήριξη. Κύριε Μπορέλ, δύο λεπτά. Δεν ξέρω αν κατάλαβα όλα όσα είπατε, αλλά πάντως βασικό μάθημα της πολιτικής είναι το νόμισμα, το σύνορο και η άμυνα. Είναι τα χαρακτηριστικά, τα βασικότερα ενός κράτους. Όχι. Τα σύνορα δεν είναι κάτι που το θαυμάζω. Εγώ νομίζω ότι είναι ουλές. Ουλές που έμειναν πάνω στο φλοιό της γης από την ιστορία και πρόοδος πάει να πει το ξεπέρασμα των σύνορων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα κλασικό παράδειγμα αυτής της υπέρβασης. Κανεί δεν υποχρεώνεται να μπει στο ευρώ. Η απόφαση προσχώρηση στο ευρώ ήταν κυρίαρχη εθνική απόφαση, κρατική απόφαση. Όποιο θέλει να κάνει αυτό το βήμα, το κάνει. Και ο οποίο θέλει να περάσει την πόρτα εξόδου, το κάνει και αυτό. Ε, εντάξει, όντω έχουν δυσκολίε κάποιε χώρε τώρα, αλλά βασική δημοκρατική ελευθερία είναι η ίδια ύπαρξη αυτή τη πολιτική κοινότητας. Αυτό οικοδομούμε. Και για πρώτη φορά στην ιστορία τη Ευρώπης αυτό δεν έχει τα θεμέλια στον πόλεμο, ίσως το ποιο είναι ο ισχυρότερο. Ούτε Ναπολεόν, Ναπολεόν ούτε Βίσμαρκ υπάρχει. Αλλά υπάρχει απλώς πολιτική βούληση και δημοκρατία. Μεγάλο κατόρθωμα και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε περήφανοι. Αν κάποιος δε δεν θέλει να συμμετάσχει σε αυτό το όραμα, υπάρχει η πόρτα της εξόδου. Θα ήθελα να σας βοηθήσω να ξανανεύετε στο τρένο τους Βρετανούς, αλλά δεν μπορώ να σας εμποδίσω. Πρόκειται για δημοκρατικό οικοδόμημα, οπότε όποιος θέλει μπορεί να αποχωρήσει. Αλλά ειλικρινά σας λέω ότι δεν μου αρέσουν τα σύνορα και στα Βαλκάνια ειδικότερα θα πρέπει να ανοίξουμε τα σύνορα. Thank you. Follow-up question, Nathan Gill. Επερώτηση από τον κύριο Nathan Gill. Α, δεν σας αρέσουν τα σύνορα, αλλά εγώ, αλλού το πήγαινε ότι είναι εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλουν, θέλουν να έχουν τα εθνικά τους σύνορα, θέλουν να διατηρήσουν την εθνική τους ταυτότητα. Αυτό που ρώτησα και δεν απαντήσατε είναι εσείς. Τι θα κάνετε από λεβάς δημοκρατικής για τους Ευρωπαίους. Δημοκρατική πολιτική, δημοκρατική νομιμοποίηση και υποστήριξη. Πώς θα το βρείτε αυτό. Ε, το καταφέρετε ή όχι. Μπορέλ. Δεν αρκεί να το θέλω να το καταφέρουμε μέσω αυτού που εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ βρίσκονται οι εκπρόσωποι, αυτοί που εκπροσωπούν δημοκρατικά τους Ευρωπαϊκού λαούς. Δεν είπα του ευρωπαϊκού λαού. Ακόμα δεν υπάρχει ευρωπαϊκό Δήμο. Έχουμε πληθώρα δήμων στην Ευρώπη. Μπορεί κανεί να είναι Ευρωπαίο χωρί να απεμπολίσει την εθνική του ταυτότητα. Ήμουν πρόεδρο Καταλανός Ισπανός Ευρωπαίος. Το είπα ως πρόεδρος και τα τρία είναι βασικά. Πολλαπλή ταυτότητα. Αυτό χτίζουμε στην Ευρώπη. Κανείς δεν εξαναγκάζεται να συμμετάσχει σε αυτό το οικοδόμημα. Αλλά είναι ό,τι καλύτερο έχει σκαρφιστεί το ανθρώπινο μυαλό. Κατά πολέμηση αυτών ε, των ταυτοτήτων έχουμε αυτές τις διαφορετικές ταυτόχρονες ε, ταυτότητες χωρίς να καταπιεστεί, χωρίς να συμπιεστεί καμία εξ αυτών. Σας ευχαριστούμε. Περνάμε στον επόμενο μιλητή για τους σοσιαλδημοκράτες, ε, Σάντσες Αμόν. Καλώ ήρθατε στο σπίτι σα, κύριε Μπορέλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο με την πυρηνική συμφωνία, σχέδιο ολοκληρωμένη κοινή δράση από Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένε Πολιτείε, Κίνα, Ρωσία, Ιράν, που υπεγράφει για να έχει τελείω μη στρατιωτικό χαρακτήρα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και το ε, έχουν πλαισιώσει και 14 ετήσια εκθέσει ε, του Οργανισμού ε, τη Διεθνού Επιτροπή Ατομική Ενέργεια. Είναι ένα παράδειγμα ευφυία αλλά και ηγεσία εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως η κυβέρνηση Τραμπ ε, που δεν θέλει το πολυμερέ αυτό πλαίσιο αποφάσισε και να αποχωρήσει από το πλαίσιο και το τορπιλίζει με μονομερεί κυρώσει κατά του Ιράκ και με εξοδαφικέ μάλιστα επιπτώσει, δυστυχώ και η και Ιράν έχουν κλιμακώσει ε, τις ε, αντιγκλήσεις και τις πιέσεις ε, και το Ιράν ξέρουμε τι κάνει και σε σχέση με τις ε, γυναίκες ε, και με την εφαρμογή του προγράμματος. Ε, πώς θα αποφύγουμε και την πυροδότηση άσχημων περιστατικών και στα στενά του γιατί το είπατε και αυτό. Πολλές ερωτήσεις μέσα σε μία και θα προσπαθήσω να απαντήσω 7 ή 8 σημεία, έτσι, τα οποία μου έρχονται στο μυαλό. Ναι, μεν αποσύρθηκαν από την ε, συμφωνία την πυρηνική είπα, όμως όλοι οι άλλοι παραμένουν ενωμένοι στο να διατηρηθεί αυτό, αυτή η συμφωνία. Δεύτερον, το Ιράν πρέπει να ε, ξαναρχίσει να εφαρμόζει πλήρως τη συμφωνία Πρέπει να αποφύγουμε δηλαδή απέναντι σε αυτή την πολιτική υψηλή πίεση από πλευρά. Ε, ε, είπα να έχουμε υψηλή αντίσταση από το Ιράν που θα μα οδηγήσει σε σύγκρουση. Εμεί ε, τηρούμε το δικό μα κομμάτι τη συμφωνία, ήραμε τι κυρώσει και προσπαθούμε να διατηρήσουμε τι εμπορικέ συναλλαγέ και τι οικονομικέ δραστηριότητε. Και επαφέ με το Ιράν έχουμε πολύ αυστηρέ διαστάσει, έχουμε πολύ αυστηρέ διατάξει και προσπαθούμε να προστατεύσουμε και τις δικές μας επιχειρήσεις. Πρέπει να συνεχίσουμε να διατηρούμε τις οικονομικές επαφές. Έχουμε και το όχι με ειδικού σκοπού για τη διευκόλυνση των πληρωμών με το ΕΡΑΝ και να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε την κατάρρευση των οικονομικών σχέσεων. Εγώ είμαι ο συντονιστής της Μικτής Επιτροπής για την πυρηνική αυτή συμφωνία και στην εντολή μου ακριβώς περιλαμβάνεται να εξασφαλίσω την εφαρμογή της συμφωνίας σε στενό συντονισμό με όλες τις πλευρές. Χρειάζεται πολιτική ενότητα μεταξύ όλων των Ευρωπαίων. Αυτή η συμφωνία ήταν το καλύτερο επίτευγμα τη διπλωματία μα και θέλω να ευχαριστήσω την κυρία ε, Μογκερίν, την κυρία Μάλπστρομ και τον κύριο Σολάνα για την εξαιρετική του δουλειά δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία αυτή να παίξουμε το γεωπολιτικό μας ρόλο. Πρέπει να μείνει ζωντανή αυτή η συμφωνία για την πρόσπιση των δικών μας συμφερόντων, της ασφάλειάς μας και για να αποφύγουμε και κάτι χειρότερο ακόμα βέβαια. Ευχαριστώ. Συμπληρωματική ερώτηση, παρακαλώ εσείς. Όχι, δεν έχετε συμπληρωματική ερώτηση. Άρα πάμε στον επόμενο ομιλητή για την ομάδα του ΕΛΚ. Αντρέι Χαλίτσκι, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να φερθώ και πάλι στην Ρωσία, η οποία είναι απειλή όχι μόνο για τις χώρες με τις οποίες συνορεύει. Ε, πολιτική παραπληροφόρηση, αποσταθεροποίησης ε, των ευρωπαϊκών κοινωνιών είναι γεγονός και θα πρέπει να αντισταθούμε σε αυτήν. Επίσης, ε, από την οικονομική σκοπιά. Αντιλαμβάνομαι ότι είστε υπέρ της διπλωματίας και όχι των κυρώσεων. Το ερώτημά μου όμως αφορά τις οικονομικές δυνατότητες. Είστε υπέρ της περαιτέρω χρηματοδότησης κάποιων έργων που υπάρχουν ήδη. Τι εργαλεία θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε στις προσπάθειες σας αυτές. Σκέφτεστε τα ΜΜΕ ή άλλα βήματα που θα μπορούσαν να αντιταχθούν σε αυτήν την πολιτική παραπληροφόρηση της Ρωσίας. Κύριε Μπορελ, δύο λεπτά. Πρέπει να επενδύσουμε πολλά για να αντιμετωπίσουμε το όπλο της παραπληροφόρησης, γιατί περί όπλου πρόκειται. Η δημοκρατία είναι ένα σύστημα που βασίζεται στην πληροφόρηση των πολιτών. Ψηφίζω με βάση τα όσα ξέρω. Εάν τα όσα ξέρω είναι λάθος, θα ε, ψηφίσω με τρόπο προκατηλημένο και ε, πλέον αμφιβάλλω για τα όσα ξέρω. Μπορώ να σας δώσω πάρα πολλά παραδείγματα. Το τελευταίο κατά τη διάρκεια των ευρωεκλογών. Πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε πολύ περισσότερο. Έχουμε τις στρατηγικές επικοινωνίες, τον πυρήνα, γρήγορη αντίδραση, αλλά είναι πολύ ευκολότερο να διασπείρει κανεί ψευδεί ειδήσει παρά να τι διαψεύσει, γιατί βεβαίω αυτές διασπείρονται πολύ πιο εύκολα. Να μπορέσει ακριβώς να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη είναι κάτι το πολύ πιο δύσκολο. Επίση, για τη Ρωσία. Δεν θέλω εδώ να φανώ ότι είμαι κατά της Ρωσίας. Είναι ένα θέμα, είναι μια χώρα η οποία μας δίνει ενέργεια, δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν υπάρχει. Πρέπει να ενισχύσουμε την Ουκρανία. Έχουμε επενδύσει 15 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία τα τελευταία χρόνια. Πολλά λεφτά. Πρέπει να γνωρίζουμε πού πάνε. Γιατί εάν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση αυτή ε, ξανατολών πρέπει να δημιουργήσουμε έναν δακτύλιο δημοκρατικών χωρών με ευημερία. Σας ευχαριστώ Έχετε και πάλι τον λόγο. Α, με ικανοποίησε αυτό το οποίο είπατε εκεί στο τέλος. Δεν θεωρείτε ότι έχουμε ένα πολύ καλό έργο που αυτή τη στιγμή δεν ε, χρησιμοποιείται. Ε, δηλαδή την Ανατολική Γειτονία. αφού βεβαίω οι γειτονικέ χώρες, η Ουκρανία και η Μολδαβία έχουν κάνει τις απαραίτητες ε, μεταρρυθμίσεις. Ε, δηλαδή το αν κατά πόσον θα αποτελέσει η ρωσική κοινωνία ένα πρότυπο. Σίγουρα, σίγουρα. Έχετε δίκιο. Τι να σας πω άλλο. Ε, δεν το έχω μελετήσει ε, ακόμη βάθος, αλλά ε, ναι, το μελετούμε. Δηλαδή η προσέγγιση Ρωσίας, Λευκορωσίας μας ανησυχεί. Ανησυχεί τα κράτη-μέλη της Βαλτικής. Και για τον Κρανία ισχύει αυτό που είπατε και θυμάμαι το 2015 που τα έλεγε η καγκελάριος Μέρκελ. Τι είναι αυτό, η τοπάθεια, ρεαλισμό και συμβασμό. Είδατε ότι ε, ήμασταν ε, λίγο πριν τον πόλεμο της Γεωργίας, παρατηρητές τις εκλογές από πλευρά όσα ο ΑΣΕ Και είδατε, το φαινόταν ότι έτσι θα γίνουν τα πράγματα και δεν έγινε τίποτα για να αναχαιριστεί. Επόμενη ερώτηση. Πινιέρο από την ΚΟΑ. Ευχαριστώ, λέει ο κύριο Πινέδα. Όταν υπεγράφει η συμφωνία του 1993, είχαμε κάποιους κάποιου του Παλαιστινίου πτώσαν στο Ισραήλ 78% και κράτησαν το υπόλοιπο 22% για να γίνει Παλαιστινικό κράτο, αλλά το Ισραήλ δεν σεβάστηκε αυτή την ε, συμφωνία, ούτε τα όσα ε, απεφάσισε ο ΙΕ και λοιπά. Και οι Παλαιστίνοι από την άλλη μεριά ε, τήρησαν αυτή την ε, συμφωνία του Όσλο και επίσης τήρησαν ότι προβλήθηκε το δίκαιο ενώ, ενώ το Ισραήλ τη ζώνη της Γάζης την, ε, την έκανε ένα νεκροταφείο και έχουμε όλα σε αυτούς τους επικισμούς, τους επίκους οι οποίοι είναι ένοπλοι και στηρίζονται από τις Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής επιτιθέμενοι στους αμυνωμένους Παλαιστινίους εκεί. Δηλαδή να είναι ε, η πρωτεύουσα των Παλαιστινίων η Ιερουσαλήμ ε, έγινε de facto πρωτεύουσα των Σιωνιστών. Θα κάνετε κάτι ούτως ώστε να ισχύσουν τα σχετικά με τους Παλαιστινίους ψηφίσματα του ΟΗΕ, Μπορέλ. Αγαπητέ βουλευτά. Γνωρίζετε ότι η ευρωπαϊκή θέση είναι το πώς θα συμβιώσουν τα δύο κράτη. Δεν ε, συμφωνούν όλοι, αλλά αυτή ήταν και ελπίζω να είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκρότηση πρώτων Παλαιστινιακού κράτους και να θωρακίζονται τα δικαιώματα των Παλαιστινίων και ταυτόχρονα ασφάλεια για το Ισραήλ. Ταυτοχρόνως και τα δύο. Και κάνουμε πολλά για τους Παλαιστινίους. Λέτε ότι δεν αρκούν, αλλά σας υπενθυμίζω ότι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει σχεδόν κάθε μέρα ένα εκατομμύριο ευρώ για να βοηθήσει την Παλαιστινιακή Αρχή. 300 εκατομμύρια ετησίως. Και αυτό από την υπογραφή της Συμφωνίας του Όσλο. Πάρα πολύ βασικό αυτό για να συνεχίσει να υπάρχει η Παλαιστινική Αρχή. Και έτσι να υπάρχει ελπίδα ότι θα υπάρξει λύση δύο κρατών. Και έχουμε αποστολή και στις δύο πλευρές. Βοηθούμε για δικαιοσύνη, για ασφάλεια κλπ. Και έχουμε και την αποστολή στην ε, Γάζα, αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα εκεί, δυστυχώς δεν είναι λειτουργική η αποστολή μας. Οπότε αν κάποιος βοηθάει τους Παλαιστινίους, ε, αυτοί είμαστε εμείς και αν κάποιος διατηρεί την ελπίδα δημιουργίας ε, Παλαιστινιακού κράτους που να συνεπάρξει συνεργά με το Ισραήλ, με εγγυήσεις και τονίζω ταυτοχρόνω το δικαίωμα ύπαρξης και ασφάλεια του Ισραήλ με το δικαίωμα των Παλαιστινίων να έχουν το κράτος τους και την πολιτική τους ε, θεσμική δομή. Ε, αυτό, αν υπάρχει κάποιος που το εξασφαλίζει, είμαστε εμείς. Όχι, δεν είμαστε κατά των Ισραηλινών απλώς. Θέλουμε να υπάρξει ειρηνική συνύπαρξη αυτών των δύο λαών που τόσο καιρό αντιπαρατίθενται. Συμπληρωματική. Ναι. Ναι. Η ανθρωπιστική βοήθεια όντως δίνεται ακόμη στην την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ευτυχώς, γιατί θα ήταν πολύ χειροτερή η κατάσταση. Αλλά χρειάζονται και άλλες κινήσεις. Πολιτική δράσεων, όχι δηλώσεων. Η κυρία Μογκυρίνη ήταν η πρωταθλήτρια των δηλώσεων που τίποτα δεν απέφεραν. Αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Άμεσα, τώρα. Τίποτε δεν δικαιολογεί την καθυστέρηση της αναγνώρισης. Έστω και αργά. Κάλλιο αργά παρά ποτέ το κάνουμε αυτό. Δεν έχει νόημα η Ευρωπαϊκή Ένωση να κλείνει το μάτι σε κάποιους που καταπατούν διεθνές δίκαιο και ψηφίσματα ε, του ΟΗΕ. Ας ισχύσει το άρθρο υπαρθμών 2 του χαρτιού για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τι λέτε. Α, δηλαδή να ακυρώσουμε τις εμπορικές συμφωνίες. Όχι. Εδώ και καιρό δεν έχουμε το Συμβούλιο σύνδεση ακριβώ για αυτό το λόγο. Άλλοι λένε να ε, γίνει εδώ και τώρα Συμβούλιο Σύνδεσης και άλλοι λένε να αναστείλουμε τις συμφωνίες. Δεν είμαι υπουργό εξωτερικών που να λέει τι πρέπει να κάνουμε εγώ. Προσπαθώ ή θα προσπαθήσω, εάν μου, με εμπιστευτείτε, να συγκεράσω τις θέσεις αυτές για να έχουμε κοινή θέση, αλλά αυτή τη στιγμή είπαμε έχουμε αντίθετες απόψεις. Αύριο, αύριο συγκαλέσατε το Συμβούλιο Σύνδεσης. Άλλοι λένε αύριο αναστήλατε τις ε, συμφωνίες. Κάθε φορά που είχαμε όλμους ε, από τη Γάζα, ή στη Γάζα τέλο πάντων, λέγανε ότι είμαι υπέρ των Ισραηλών και το αντίστροφο λέγαν ότι είμαι επικίνδυνος και είμαι κατά των Ισραηλινών. Άρα έχουμε το μαύρο και το άσπρο και θα πρέπει να τα συγκεράσουμε για να βρεθεί μια θέση. Ευχαριστούμε κύριε Μπορέλ, ο πρόεδρος. Κάτι πήρε για τους σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε Μπορέλ που μας είπατε σήμερα το πώς βλέπετε τις διάφορες προκλήσεις ε, που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μετανάστευση και η ένταξη πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα τα επόμενα χρόνια παρά τις δηλώσεις κάποιων κρατών μελών ότι το κλείσιμο των συνόρων είναι δυνατό. Όμως, πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να σταματήσουν οι τραγωδίες στη Μεσόγειο και να φροντίσουμε η μετανάστευση να γίνεται με τρόπο έφτακτο και ασφαλή. και επιπλέον η σχέση μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής σχέσης είναι πάρα πολύ σημαντική. Τι γίνεται λοιπόν για να αντιμετωπιστούν οι αιτίες της μετανάστευσης και πώς ε, σκοπεύετε να ενισχύσετε τη συνεργασία με τις ε, χώρες διελευσής. Κύριε Μπορέλ, δύο λεπτά. Νομίζω πως ε, η μετανάστευση πρέπει να ενσωματωθεί πλήρω στην εξωτερική πολιτική. Δεν είναι στο χρονοδιαγραμμά μου, αλλά είναι κιόλα. Αλλά δεν θα λύσουμε το πρόβλημα αυτό χωρίς ε, συμφωνίες ε, με τις χώρες προέλευση και διέλευση. Αν πάτε στη Σενεγάλη θα δείτε πως η Ευρώπη είναι μαγνήτης, μαγνήτης στις Εάν ε, δεν μπορέσουμε να διακρίνουμε μεταξύ όσων ζητούν άσυλο και ατόμων που δεν ε, έχουν δικαίωμα διεθνούς προστασίας, πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε συμφωνίες με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης για να υπάρχει μια άμεση αντίδραση. Γνωρίζετε τι συμβαίνει σήμερα στα νησιά στην Ελλάδα. Αυξάνεται. Αυξάνονται οι αφήξεις. Τους τελευταίους δύο μήνες έχει αυξηθεί ε, μιλάμε για 20.000 άτομα σχεδόν. Οι περισσότεροι είναι Αυγανοί, δεν είναι Σύριοι. Ε, τι θα τους κάνουμε. Δεν μπορούμε να λέμε ότι θα κάνουμε μια τέτοια συμφωνία και μετά να μην μπορούμε επί τόπου να κάνουμε αυτήν την διάκριση και να τους αφήνουμε στις παραλίες γιατί δεν ξέρουμε τι να τους κάνουμε. η μεταναστευτική πολιτική είναι πολύπλευρη. Για πολύ επίπεδη. αλλά το πρώτο το οποίο πρέπει να γίνει είναι να συμφωνήσουμε με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης για να γίνει ε, έφτακτη. Και ε, αφενός ε, έχουμε κατά νου την κορύφωση αυτή του 2015-16 που πρόκειται για πρόσφυγες 1,5 εκατομμύριο Τώρα οι αριθμοί δεν είναι 1,5 εκατομμύριο. Μιλάμε για 20-30 Για ολόκληρη την περιοχή. Αυτό δεν είναι εισβολή, αλλά προσοχή. Και σβήνει το μικρόφωνο του κυρίου Μπορέλ. Σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό πάλι κυρία Κατυπήρη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την Προεδρία σας και είμαι σίγουρη ότι στο μέλλον θα έχουμε και περισσότερο χρόνο με τον κύριο Μπορέλ για να το συζητήσουμε. Πώς ε, μπορούν, Πώς βλέπετε να εφαρμοστούν οι δομές που έχουν συμφωνηθεί στο Συμβουλίο για να διασφαλίσετε ότι θα υπάρξουν οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης οι οποίες θα αποποινικοποιηθούν στη Μεσόγειο σε συνεργασία με τις προσπάθειες των κρατών μελών για να σώσουμε ζωές και να καταπολεμήσουμε την παράνομη διακίνηση. Σας ευχαριστώ κύριος Μπορέλ. Κύριε Βουλευτά, αν με εμπιστευτείτε. Ελπίζω να έχω την τύχη να συνεχίσω τη συζήτηση για το θέμα αυτό, γιατί με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Τα δύο τελευταία καλοκαίρια ω ε, πρόεδρο εξωτερικών τη Ισπανία τα πέρασα με το τηλέφωνο στα αυτή, προσπαθώντα να βρω μία λύση με αυτά τα σκάφη με 200 άτομα στη Μεσόγειο που δεν τα ήθελε κανένα. 200 άτομα και δεν τα ήθελε κανεί. Η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί τέτοιες καταστάσεις. Δεν μπορούμε να δεχθούμε κάθε καλοκαίρι να συζητούμε ξανά και ξανά τι θα κάνουμε με 200 άτομα. Πρέπει να έχουμε μια συμφωνία που αυτόματα να μας επιτρέπει να ε, αφήνουμε αυτούς τους ανθρώπους να βγουν στη στεριά και μετά να δούμε τι θα τους κάνουμε. Δεν είναι πρόβλημα για την Ευρώπη. Το πρόβλημα είναι ότι είμαστε απρόθυμοι να καταλήξουμε σε συμφωνία. Το είπα και το ξαναλέω. Πρέπει να γίνουν σεβαστές ιδιαιτερότητες, διαφορετική ιδιοσυγκρασία της κάθε χώρας ε, σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση. Δεν τα αντιλαμβανόμαστε με τα ίδια τρόπο. Όμως, ως πολιτισμός, γιατί μιλάμε καθημερινά για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν μπορούμε κάθε Αύγουστο να καθόμαστε στι οθόνε τη τηλεόραση ή ε, υπουργοί εξωτερικών να είμαστε με ένα τηλέφωνο στα αυτιά προσπαθώντα να συνοηθούμε ότι θα κάνουμε 200 άτομα. Στην Κολομβία, ξέρετε, έχουν 3 εκατομμύρια από τη Βενεζουέλα. 3 εκατομμύρια από τη Βενεζουέλα. Τι θα γινόταν στην Ισπανία αν έρχονταν 3 εκατομμύρια Πορτογάλοι, μπορείτε να το φανταστείτε, μας φοβίζουν 200 άτομα. Ευχαριστούμε. Περνάμε στην κυρία Γκριγορόβα από τους Πράσινους. Ευχαριστώ και καλώς ήρθατε κύριε Μπορέλ. Με μεγάλη μου χαρά άκουσα ότι αναγνωρίσατε την παραπληροφόρηση ως πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ είναι κάποιες περαιτέρω διευκρινήσεις. Λοιπόν, τι συγκεκριμένα μέτρα θα λάβετε για να καταπολεμήσετε την παραπληροφόρηση και την παρέμβαση στις εκλογές και μαζί με αυτό πώς θα εγγυηθείτε την ελευθερία λόγου και θα προλάβετε την λογοκρισία στις εκλογές, στο διαδίκτυο. Ε, επίσης, ε, θα ήθελα να μάθω τι θα κάνετε για τις πωλήσει όπλων και για την κοινή θέση ε, να σας ρωτήσω λοιπόν, σκοπεύετε να ενισχύσετε τον έλεγχο όπλων ε, των, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μετατραπεί σε κοινωτικό δίκαιο. Σας ευχαριστώ κύριε Μπορέλ για δύο λεπτά. Και πάλι δύο ερωτήσεις σε μία. Κοιτάξτε, για τις εξαγωγές όπλων. Έχουμε μια κοινή θέση από το 2008, η οποία είναι νομικά δεσμευτική για τα κράτη-μέλη. Εφαρμόζεται βεβαίως ε, με την ευθύνη των κρατών μελών. Η κοινή αυτή θέση απαιτεί 8 κριτήρια αξιολόγησης που πρέπει να ακολουθήσει κάθε κράτος μέλος για να εγκρίνει μια εξαγωγή όπλων, αλλά μπορεί να αρνηθεί μια εξαγωγική άδεια εάν πρέπει εάν βλέπει ότι υπάρχει σαφής κίνδυνος για παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. αυτή είναι οι κανόνες. Δυστυχώς, η Κομισιόν, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, εμείς δηλαδή τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, δεν έχουμε έντολη να παρακολουθούμε τις αποφάσεις των κρατών μελών για τις άδειες όπλων. Δεν έχουμε τέτοια εντολή, αλλά δώστε την. Αλλά μην μας ζητάτε να εφαρμόσουμε ε, δράσεις ε, για τις οποίες δεν έχουμε αρμοδιότητα. Τελική απόφαση είναι στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Και σας υπενθυμίζω ότι στο θέμα αυτό απαιτείται ομοφωνία και υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ των κρατών για το θέμα αυτό. Και απαιτείται ομοφωνία. Και οπωσδήποτε είναι ε, αδύνατο να γίνει με την ομοφωνία. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, να επαναδιαπραγματευτούμε τη συμφωνία του 2008 απαιτώντας πρώτα απ' όλα ανταλλαγή πληροφοριών. Πρέπει να ξέρουμε το τι κάνει κάθε χώρα. Σε ποιον, με ποιον και όπως κάνουν μερικές χώρες ε, το πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα όπλα. Σας ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση. Ε, συγγνώμη για το ότι η ερώτησή μου σας έκανε να αποφύγετε το θέμα της ε, παραπληροφόρησης. Έχω και άλλη μια ερώτηση. Η θέση για την οποία είστε υποψηφίος ε, είναι οπωσδήποτε κάτι το πάρα πολύ σημαντικό ότι πείτε θα εκπροσωπεί 500 εκατομμύρια Ευρωπαίων. Θα πρέπει λοιπόν να αποτελείται ένα πρότυπο. Δεδομένου του ιστορικού σας με συγκρόμνα συμφέροντα, παρέτηση από το Πανεπιστήμιο και ένα πρόστιμο 2.000 ευρώ για εσωτερική πληροφόρηση στο χρηματιστήριο θα σκεφτείτε να πουλήσετε όλες σας συμμετοχές για να μην έχετε άλλα τέτοια μπλεξίματα. Κύριε Μπορέλ. Κοιτάξτε, ήδη σας εξήγησα το ζήτημα αυτών των εμπιστευτικών πληροφοριών αλλά σας ευχαριστώ που το ξαναρωτάτε γιατί μου δίνετε την ευκαιρία και εγώ να τα ξαναπώ. Κάποιος ο οποίος κάτι κάνει για το 7% του χαρτοφυλακίου του μένει το υπόλοιπο 93% και χάνει για κάτι που κάνει 300.000 ευρώ, ε, να τα χάσει όλα, είναι τελείως ηλίθιο. Αν εγώ έκανα κάτι τέτοιο θα ήμουν και εγώ τελείως ηλίθιος. Το 7% ρισκάρεις και χάνει το 93%. Ποτέ θα έκανα κάτι τέτοιο να παραβώ την υποχρέωση της εμπιστευτικότητας και νομίζω ότι είναι λογικό αυτό το οποίο σας λέω. Μήπως και δεν παρευρίασα το καθήκον εμπιστοσύνη. Δεύτερον, όσον αφορά την... Α, λέτε για μετοχές. Ναι. Στην ε, νομική επιτροπή υπήρχε ένα θέμα. Ότι εγώ είχα 12.000 ευρώ μετοχές της ε, Ιμπερδρόλα. Εάν αυτό σα ενοχλεί, τότε αύριο θα ζητήσω να πολιθούν. Κανένα πρόβλημα. Με τίποτα. Αύριο να λυθεί κιόλα. Τώρα, όσον αφορά την παραπληροφόρηση, τον σταματά ο πρόεδρο γιατί περίβει το χρονικό όριο. Ευχαριστούμε κύριε Μπορέλ. Ο επόμενο. Χαβιέρ Νάρτ από του Φιλελευθέρου. Κύριε Μπορέλ, καλώ ορίσατε εδώ στο Κοινοβούλιο. Μιλήσατε για την ασφάλεια όσον αφορά τα νότια σύνορά μας για την, με την Βόρεια Αφρική. Εκεί ε, άμεσα ε, υπάρχουν επιπτώσεις από το τι γίνεται σε Σαχάρα, σε Σαχέλ, άρα η ασφάλεια της περιοχής εκείνης ε, είναι η ασφάλεια δική μας. Υπάρχει επομένως εδώ το θέμα ανάπτυξη, σταθερότητα, ασφάλεια, τρίγωνο. Και τα πράγματα Ολλάνδοι και γίνονται πιο καυτά εκεί με κάθε έννοια. Δηλαδή έχουμε κάποιες ιστορικές συγκρούσεις που έχουν την ρίζα τους σε Ισλαμισμό και τρομοκρατία. Εσείς ως είπατος εκπρόσωπος, τι θα κάνετε για αυτό το πρόβλημα που πρόκειται για αυτό το θέμα σταθερότητας, ανάπτυξης, ε, ασφάλειας και αυτό το τρίγωνο. Έχετε δύο λεπτά κύριε Μπορέκη. Ναι, σωστά το λέτε. Πρόκειται για ένα τρίγωνο και έχουμε κλίμα, τρομοκρατία επίσης και το τρίγωνο δεν θα αντιμετωπιστεί κάνοντας κάτι μόνο για με πλευρές. 50% είναι κάτω κατόφλητες στόχες εκεί. Το 1 τρίτο των σχολείων στην Πουρκίνα Φάσο έχουν κλείσει η ασφάλεια. Αυξάνεται παρά τις προσπάθειες που έχουμε καταβάλει προς το αντίθετο είμαστε ο βασικός δωρητής. Και τα τελευταία 7 χρόνια έχουμε χορηγήσει σχεδόν 4 δις ευρώ στο Σαχέλ. Αν όμως πραγματικά θεωρούμε ότι είναι δυνατόν να υπάρξει ε, κάτι, κάποιο μέτρο για 5 εκατομμύρια τετραγωνικών χιλιόμετρων, 10 φορές όσο στην Ισπανία και έχουμε εκεί πέρα 200 εκατομμύρια κατοίκων και ότι μπορούμε κάτι να κάνουμε με 300 χωροφύλακες και συνοριοφύλακες για κάποια σύνορα που δεν υπάρχουν, ε, αυτό δεν θα είναι ρεαλιστικό και βέβαια το να μην ε, επενδύουμε στο Σαχέλ κοστίζει πάρα πολύ, άρα θα πρέπει κάτι να κάνουμε και θα πρέπει επομένως να επενδύσουμε εκεί από πάσης απόψεως. Ιδάλλως, Ιδάλλως. ξέρετε που πρέπει να αρχίσουμε να αρχίσουμε με την χειραφέτηση της γυναίκας. Πηγαίνετε κάπου στον Ήγηρα, σε ένα μευτήριο, να δείτε τι γίνεται. Θα συνειδητοποιήσετε ότι υπάρχουν κάποιες κοπέλες που έχουν 7-8 παιδιά με στη φτώχεια. Ε, έτσι καταλαβαίνετε γιατί έχει ξεφύγει το δημογραφικό και έχει, ε, είναι προβληματική ο κοινωνικός ε, ιστός. Άρα χρειάζεται και στο πολιτιστικό ε, μέτωπο να προσπαθήσουμε. Δεν γίνεται αυτό με διάταγμα, δεν γίνεται με μια οδηγία. Να πούμε ότι αύριο αλλάζει η νοοτροπία. τίποτα δεν θα αλλάξει. Όλα θα μείνουν ίδια. Θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο σε κάθε επίπεδο και το κόστος του να μην το κάνουμε θα είναι τεράστιο για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Επερώτηση, κ. Σνάρντ, Μιλήσατε για δημογραφική ανάπτυξη για τον Νίγηρα. Είναι πρωταθλητέ στον κόσμο στον Νίγηρα. Αλλά εγώ είπα για δύο άλλε διαφορετικέ πολιτικέ. Την Πουρκίνα Φάσο, που είναι χώρα συγκροτημένη και άλλη μία που δεν υπάρχει ουσιαστικά, που είναι το Μαλί, δεν υπάρχει εκεί κράτο. Και εκεί τα πράγματα χειροτέρεψαν παρά την ε, στρατιωτική εκπαίδευση, παρά την οικονομική βοήθεια. Εσείς τι θα κάνατε. Ε, εν ώψη αυτής της επένδυσης που δεν αποδίδει. Πριν από τέσσερα χρόνια είχαμε την Συμφωνία Ειρήνευση στο Μαλί. Και πολύ λίγα με το πρώτο έχουν γίνει από τότε. Είναι χώρα πολύ σημαντική. Επηρεάζει φυσικά το τι γίνεται στην Μπουρκίνα Φάσο. Ακριβώς. Πρόκειται για ένα σταυροδρόμι εθνοτήτων, πολιτικών, ε, θρησκευτικών διαφορετικών, ε, διάφορη διαπλοκή αντίθετων συμφερόντων και υπήρχαν και συγκρούσεις πολύ πριν την Ισλαμική τρομοκρατία. Οπότε έτσι μεταδίδεται η ανασφάλεια και αλλού. Κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να εμπλακούμε περισσότερο, να στείλουμε περισσότερες ειρνευτικές αποστολές για να Βοηθήσουν να φτιαχτεί το κράτος. Δεν το καταφέραμε στο Σαχέλ, αυτό είναι το πρόβλημα. Άμυνα, ασφάλεια, αστυνομία, ό,τι είχε αφήσει η επικοινωνία μόνο αυτά λειτουργούν. Αλλά από πλευράς παροχής κρατικών υπηρεσιών δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει ένα κράτος πολύ τη βία. Ε, αυτό τίποτα δεν έγινε σε αυτό το μέτωπο. Εκεί πρέπει να προσπαθήσουμε. Να υπάρχουν κάποιες σύγχρονες δομές και να μην συνεχίζουν να υπάρχουν οι αρχέτυπες, οι παλιές δομές, οι προ της απεικιοκρατίας. Thank you, Mr. Borel. We come to the final... Ευχαριστώ, κύριε Μπορέλ. Τελευταίος ομιλητής, Μίχαλ Γκάλερ, από το ΕΛΚ. Η συζήτηση εδώ πέρα με παρακίνησε να κάνω άλλη μία ερώτηση για την Κούβα. Λέτε ότι όλοι πηγαίνουν εκεί. Η αλήθεια είναι σχεδόν όλοι, αλλά όχι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα δεσμευτείτε να μας ε, στηρίξετε για να μπορέσουμε να πάμε μια αποστολή με τη σύντηση που θέλουμε εμείς και να μιλήσουμε σε όποιον θέλουμε εμείς σκοπεύεται να υπάρξει ε, μια ευρωπαϊκή πολιτική με οδικό χάρτη για ελεύθερες εκλογές στην Κούβα. Γιατί τα στηρίζουμε αυτά στην Ουκρανία και αλλού, στην Τουρκία, στην Τινησία, στη Βενεζουέλα και οπουδήποτε στην Αφρική, αλλά απογοητεύουμε τους Κουβανούς. Οι Κουβανοί ούτε με τον Μπατίστα είχαν εκλογές, ούτε με τους Κάστρο δεν αξίζουν ελεύθερες εκλογές. Έχετε κάποιο επιχείρημα ε, για να στηρίζετε αυτούς τους πολιτικούς ε, δεινόσαυρους. για να αρνείστε τα θεμελιώδη δημοκρατικά του δικαιώματα και ελευθερίες. Κύριε Μπορελ, δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γκάλερ. Νομίζω ότι... Νομίζω πως μάλλον υπήρχε κάποιο πρόβλημα στην διερμηνία. Δεν είπα ότι πάνε όλοι στην Κούβα πλην του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είπα σχεδόν όλοι εκτός από τον βασιλιά της Ισπανίας. Δεν είπα τίποτα για Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν ξέρω τι θέλετε να κάνετε, αλλά το γεγονός είναι πως έχουν πάει όλοι στην Κούβα πλην τη Ισπανίας. Και πιστέψτε με, έχουμε ε, σοβαρούς ιστορικούς δεσμούς με την Κούβα. Και πολλοί είναι ισπανική καταγωγής. Οπότε δεν λέω τίποτα υπέρ ε, του ότι η Κούβα είναι δημοκρατική χώρα λοιπά, Γιατί οπωσδήποτε δεν είναι. Οπωσδήποτε δεν είναι. Και πρέπει ακριβώς να προσπαθήσουμε ε, να γίνει η κοινωνία πιο ελεύθερη. Και ακριβώς θα πρέπει να έχουμε σχέσεις, να έχουμε κάποιο σημείο επαφής. Δηλαδή το να κλείνουμε την πόρτα και να τους μπλοκάρουμε ε, δεν ήταν καθόλου χρήσιμο και επιτρέψατε μου. Εάν θέλετε να μιλήσουμε για ανθρώπους που δεν ε, γίνεται σεβαστή η δημοκρατική της ελευθερία, υπάρχουν χώρες πιο κοντινές στην Ευρώπη. Δεν δικαιολογεί αυτό τίποτα. Όχι, όχι. Εντάξει, ε, όπως λέμε, δεν ε, δικαιολογεί η πανούκλα τη χολέρα, αλλά εντάξει. δεν έχει ε, υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Ούτε η Κούβα είναι μια δημοκρατική ανομαλία ή αδημοκρατική ανομαλία. Τουλάχιστον δεν υπάρχουν καταδίκες ε, θανάτου ούτε σταυρώσεις. Έχετε ένα λεπτό κύριε Γκάλερα. Ναι, επανέρχομαι στην ερώτηση που ήθελα να κάνω αρχικά την ειδική σχέση ε, κομισιών και Κοινοβουλίου θα, έχουμε, θα είστε εταίρος ε, διακυβερνητικός ή της κοινοτικής μεθόδου. Και ποια θα είναι η συνεργασία σας με το Κοινοβούλιο για την διαμόρφωση της στρατηγικής αλλά και πρακτικά ε, τα επιτυχημένα παραδείγματα π.χ. από Ουάσιγκτον και Χάγη αποδεικνύουν την χρησιμότητα της ε, συνεργασίας των γραφείων και των αντιπροσωπιών μας. Προτείνεται λοιπόν να ανοιχθούν τέτοια γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε Νέα Υόρκη, Αντίσα Μπέμπα και Τζακάρτα, αντίστοιχα στα Ηνωμένα Έθνη, στην Αφρικανική Ένωση και στο Ναζίαν. Κύριε Μπορέλ, ο Παναγία μου. I, cannot ensure you that. I don't know what you are talking. Δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Ε, δηλαδή, δεν ξέρω γιατί πράγμα μου μιλάτε. Ειλικρινά. Μπορείτε να είστε κάπως πιο συγκεκριμένος. Δηλαδή, ακριβείς ήσασταν. Ε, αντιλήφθηκα την ερώτηση. Ε, απάντηση δεν έχω. Okay. Θα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους ε, βουλευτές αλλά και τον ε, είπα το πρόσωπο. Θα δώσω τώρα τον λόγο και πάλι στον κύριο Μπορέλ για μια σύντομη δήλωση 5 λεπτών. Έχετε τον λόγο. Να πιω λίγο καφεδάκι. Ευχαριστώ. Ναι, είναι βεβαίως λέει ο πρόεδρος. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Θα Σα ευχαριστήσω όλους για τις σημαντικές ερωτήσεις, για την άριστη συζήτηση που κατέδειξε πόσο κινούμεθα στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά και πόσες διαφορές. Επιτρέψτε μου κάποιες τελικές σκέψεις. Να, να, να σας τα πω αυτά για να δείτε ότι τα ξέρω και τα Ιταλικά. First, it seems to me... Πρώτα απ' όλα, πρώτα σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική και αφού σας άκουσα όλους και αφού είδα πώς προετοιμάσατε, πόσο προσεκτικά προετοιμάσατε αυτή την ακρόαση, έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τρία προβλήματα έχει να αντιμετωπίσει. Ταυτότητα, τοποθέτηση στον κόσμο και μέθοδο. Ταυτότητα καταρχάς. Ε, εξακολουθούμε να διστάζουμε για το κατά πόσο είμαστε ένας παγκόσμιος πρωταγωνιστής που χρησιμοποιεί όλα τα μέσα ισχύω ήπια και μη ή όχι. Εγώ νομίζω ότι ακόμη δεν ε, δρούμε όπως θα έπρεπε και θα έπρεπε να δείξουμε πυγμή πολύ περισσότερο. Δεύτερον, η τοποθέτησή μας ε, κοινή θέση δυσκολευόμαστε να έχουμε απέναντι στις μεγάλες ε, δυνάμεις του κόσμου, ε, τη Δύση, στην Κίνα, τη Ρωσία και με τις ε, μεσές δυνάμεις, με κάποιες συγκεκριμένες περιφέρειες και θέματα μπορεί να είμαστε καλύτερα, αλλά με τις μεγάλες, με τις υπερδυνάμεις αποφεύγουμε τη συζήτηση ή οθετούμε μια τεχνοκρατική προσέγγιση με τις χιλιάδες ε, τα ανακοινοθέντα. Τρίτον, το πρόβλημα η μέθοδος. Το θεσμικό σύστημα της ΕΕΔ και της Κομισιόν εξ όσων εγώ κατανοώ τα πράγματα και δεν θέλω να σκίσω σε κανέναν κριτική, είναι policy light process heavy. Και νομίζω ότι θα πρέπει να εργαστούμε για να προσφέρουμε πραγματική προστιθέμενη αξία σε αυτά που θέλουν και χρειάζονται τα κράτη. Βλέπουμε μία τάση επανεθνικοποίησης, επανακρατικοποίησης της εξωτερικής πολιτικής πίσω στις πρωτεύουσες, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα κράτη-μέλη. Και ποιος είναι πιο έτοιμος να αναλάβει δράση πάντα, ξέρουμε και καταλαβαίνουμε τι εννοώ. Μπορεί κάποιος να μην το αρέσει, όμως ε, νομίζω αυτό δείχνει την ανάγκη να είναι πιο προσαρμοσμένο ε, το ευρωπαϊκό σύστημα, να μην υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις και γραφειοκρατία. Να έχουμε μια βαθύτερη, πιο σωστή στρατηγική ανάλυση, κάτι που δεν κάνουμε σε επαρκή βαθμό. Θα πρέπει δε να επανακτήσουμε την αίσθηση της ανάληψης πρωτοβουλίας και δράσης. Μπορεί κανείς να με ρωτήσει ε, τι ε, μπορεί να περιμένει από μένα. Ακριβώς αυτό να περιμένει. Την ανάκτηση πρωτοβουλίας και δράσης. Δεν μπορώ να είμαι παντού, όμως υπάρχουν 28 ή τέλο πάντων 28 Υπουργοί Εξωτερικών που μπορούν να με βοηθήσουν. Μπορούν να βοηθήσουν τον υπατοεκπρόσωπο μπορούν και αυτοί να ταξιδέψουν, να ε, βοηθήσουν ε, σε συγκεκριμένα θέματα, γιατί μπορεί κάποιες χώρες να τα ξέρουν καλύτερα από κάποιες άλλες ορισμένα θέματα. Και έτσι θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη οικειοποίηση ε, της ευρωπαϊκής πολιτικής η Ένωση και θα σας, βοηθήσω, θα σας ζητήσω να βοηθήσετε και εσείς στο να έχουμε πιο πολλά ποιοτικά στρατηγικά έγγραφα που θα αναφέρουν και τις πολιτικές επιπτώσεις. Γιατί κάποιος είπε ότι πρέπει να έχουμε μια πολιτική θεώρηση. Αυτό θέλουμε στην Ευρώπη, αλλά και μεταξύ Ευρώπης και πρωτεύουσών. Εμείς δεν θα κάνουμε κάτι που δεν θα το θέλουν οι πρωτεύουσε και οι κυβερνήσεις πρέπει να καταλάβουν ότι εμείς αυτό που προσφέρουμε είναι προστιθέμενη αξία, κοινή σκέψη, συγκέντρωση πόρων και δυνατοτήτων. Ξέρω με βουλευτές, η εξωτερική πολιτική ουσιαστικά δείχνει έναν τρόπο αντίληψης ε, του κόσμου και είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία και οι μας παραδόσεις είναι διαφορετικές. Δεν κατανοούμε με τον ίδιο τρόπο τις σχέσεις με τη ΣΥΠΑ, οι Πολωνοί, οι Ισπανοί, όχι. Όμως, έχουμε το κοινό αυτό όραμα για τον κόσμο. Γι' αυτό είμαστε μαζί. Αντιλαμβανόμαστε με τον ίδιο τρόπο τον κόσμο και την ανάγκη να προστατεύσουμε τον πολιτισμό μας. Πολιτισμό το λέμε, γιατί οι Ευρωπαίοι είμαστε πολιτισμός, δημοκρατία, αλληλεγγύη, ευημερία. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις αντιπροσωπείες της Ένωσης με πολύ καλύτερο τρόπο. Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων είναι φορέας λήψος αποφάσεων, σας πενθυμίζω, που πρέπει να προσφέρει καθοδήγηση, να κάνει διάλογο, αλλά να καταλήγει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, σε κοινέ δράσεις. Είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και το κάθε να πηγαίνω εκεί και να καταθέτω τα σημαντικότερα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό προνόμιο και θέλω μαζί σας να το κάνω αυτό. Και τέλος, αυτό Sarò lieto di lavorare in stretta collaborazione con il Parlamento. Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί είμαι πεπισμένο για τι δυνατότητε τη κοινοβουλευτική ε, διπλωματία. διότι γνωρίζω καλά ότι τα ψηφίσματά σα, η διαμεσολάβησή σα, οι αποστολέ ε, παρατηρητών σε εκλογέ έχουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για τη διαμόρφωση τη εξωτερική Ευρωπαϊκή Πολιτική και την αξιοπιστία της.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 σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τελευταία σας αυτή δήλωση. Σας ευχαριστώ που απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ τελειώνει η ακρόαση. Ε, καλό σας βράδυ εύχομαι και μπράβο σας κύριε Μπορέλ.